Dear colleagues, good την πρώτη συνεδρίασή μας μετά τις θερινές λέει ο Πρόεδρος. Και ελπίζω όλοι να περάσατε υπέροχα κατά αυτές τις διακοπές και γυρίσατε γεμάτη σφρίγους, γεμάτη ενέργεια και έτσι θα καταστεί δυνατό να μπορέσουμε να εργαστούμε τώρα αμέσως. Οπότε, καλώς ορίσατε και πάλι. Πρώτο σημείο, η έγκριση της ημερησίας διατάξεως. Και σας ενημερώνω ότι έχουμε κάποιες αλλαγές στην ημερησία διάταξη. Πρώτα πρώτα το θέμα υπαριθμών 19 πρέπει να συζητηθεί μετά το σημείο υπαριθμών 3. Το σημείο 4 θα συζητηθεί μετά το 13. Το 5 θα συζητηθεί μετά το 23. Τα 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 25 και 26 αναβάλλονται. Όμως σας προτείνω να εξετάσουμε την δήλωση των οικονομικών συμφερόντων του κ. Τζούλια Κίγκ. Να το συζητήσουμε λέγω μετά το σημείο 24. Έχετε κάποιες ενστάσεις για αυτά, όχι από ό,τι βλέπω. Οπότε θα πρέπει να σας πω ε, ευθύς εξ αρχής ότι έχουμε μία καινούρια τεχνική της, ε, ε της ε, αποτύπωσης σε, ταινία τη συνεδρίασής μας και γίνεται πειραματικά σήμερα μία ε, τέτοια βιντεοσκόπηση ε, οπότε σε ακτίνα των 60 μοιρών θα ε, βιντεοσκοπηθεί η συνεδρίασή μας στην είπαμε πειραματικού χαρακτήρα, δεν πρόκειται να μεταδοθεί κάπου. Τέλο πάντων, προχωρούμε τώρα και πάμε στο σημείο υπαριθμών 2, οι ανακοινώσει του Προέδρου. Επιτρέψτε μου να σα πω το εξή. Ίσως γνωρίζετε ότι από τότε που είχαμε το δημοψήφισμα σήμερα με το οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο επιθυμεί να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαμε μια σειρά επιθέσεων ξενοφοβικών και ρατσιστικών κατά πολιτών της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, οι οποίοι ε, τελείως ε, νόμιμα κινούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και βέβαια κορυφώθηκαν τα γεγονότα με την δολοφονία της ε, Τζο Κόξ, η οποία ήταν υποψήφια βουλευτής, βουλευτής μάλλον και είχε διατελέσει και συνεργάτης βουλευτού εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο Χάρλογκ αυτό, στο Έσεξ αυτή η βάρβαρη επίθεση και επίση είχαμε και την ε, ε, ανθρωποκτονία του Αρκάντη Γιούσβικ, ενός ε, Πολωνού. Γνωρίζετε βέβαια ότι εμεί πάντοτε δίνουμε τον αγώνα για τα νόμιμα δικαιώματα και για την δικαιοσύνη και ο κύριος Γιούσβικ διέπραξε το έγκλημα να μιλήσει τη γλώσσα τα απορρονικά. Οπότε δεν μπορούμε παρά να στείλουμε τα συλληπιτηριά μας προς ε, την οικογένεια και τους φίλους του Βερκάντη Γιούσβικ. Παρακαλώ να τηρηθεί ενός λεπτού συγγύη στη μνήμη του.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 That's all for the announcements. Now, ναι. approval of the minutes, if there is no objection... Αν δεν έχετε καμία ένταση, επομένως τότε θα θεωρηθεί ότι εγκρίνεται τα πρακτικά των συνεδριάσεων που συνέβαινε σήμερα σε διάταξη, δηλαδή 11 και 12 Ιουλίου 2016 και Ιουνίου 2016, ε, θα θεωρηθούν εγκεκριμένα λίγο και Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε με το σημείο υπαριθμών 19. Το 19. Έκθεση πεπραγμένων όσον αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Προϋπολογισμών ε, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Μας αναφέρει η συνάδελφος θα λάβει το, το λόγο, αλλά και η κύρια Χάνιμπολ. Γιατί αυτές οι δύο συνάδελφοι, η κυρία Κάτσια πρώτη, ε, είχε και εκείνη παραστήσει συνεδρίες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και έχουμε αυτές τις ε, σημειώσεις από τα πεπραγμένα εκεί, τα οποία είναι αρκετά εκτεταμένα και η Καρίν τα κάλυψε όλα όσα συζητήθηκαν. Εγώ έχω λίγα να προσθέσω ότι δηλαδή πρόκειται για την ε, πρώτη συνάντηση. Οπότε και οι πρόσωποι τη Επιτροπή μα παρέθησαν εκεί, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και εγώ ε, και η συνάδελφο ε, πήγαμε μαζί ε, και παρέστημα στην συνεδρίαση και πρόκειτο για την πρώτη σχετική συνεδρίαση. Οπότε θεωρήσαμε ότι το καλύτερο είναι και οι δύο να παραστούμε εκεί ούτως ώστε να μπορέσουμε να ακούσουμε ποια είναι τα θέματα, να είμαστε προετοιμασμένες και έτσι να μπορέσουμε να έχουμε μια σωστή αφετηρία για να συνεχίσουμε το έργο μας αργότερα. Οι ληφθείς σας αποφάσεις αναφέρονται σε αυτό το σχετικό σημείωμα και έχουμε επίσης δύο ζητήματα για τα οποία πρέπει να σας εξηγήσω δύο πράγματα. Πρώτα-πρώτα όσον αφορά την ε, σύσταση ότι η απόσπαση θα συνεχίσει να ισχύει για κάποιους υπαλλήλου, αυτοί που έχουν οριστεί ως πρόεδροι, ως πρόεδροι του, του ε, δευτεροβάθμιου ε, δικαιοδοτικού οργάνου. Οπότε είπαμε ότι έχουμε κάποιες προκαταρτικές παρατηρήσεις από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και αφορούν το πώς οι υπάλληλοι ορίζονται σε αυτό το δικαιοδοτικό δευτεροβάθμιο όργανο και επί τη βάση αυτών των παρατηρήσεων λοιπόν του Ελεκτικού Συνεδρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι τουλάχιστον οι διοικητικοί υπάλληλοι της ε, υπηρεσίας ε, είπαν ότι μπορούμε να συνεχίσουμε αυτόν τον τρόπο και μπορούμε επίσης να επιφέρουμε τις αλλαγές που έχουν η προτείνει. Και οι μερικοί εγώ είπαμε ότι οι προτινόμενες αλλαγές δεν καλύπτουν αυτά τα οποία έχει παρατηρήσει το ελληνικό συνέδριο διότι είπαμε ότι οι υπάλληλοι οι οποίοι εργάζονται στην υπηρεσία πνευματικής ιδιοκτησίας προβλέπεται να ε, να, να επικουρούνται από, από, άλλα, από άλλους υπαλλήλους στο δεύτερο βάθμιο αυτό όργανο. Εμείς είπαμε ότι είμαστε υπέρ μιας τέτοιας ε, αποφάσεως γιατί νομίζουμε ότι έτσι θα καλύψουμε το ελεγκτικό συνέδριο. Αλλά επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αναλύσει το πώς μπορούμε ε, αυτή τη διαδικασία να την ε, θωρακίσουμε τόσο ώστε να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις σε σχέση με την αντικειμενικότητα των μελών αυτού του οργάνου. Αντικειμενικότητες λοιπόν και αμεροληψία. Να μην υπάρχει καμία σκιά αμφιβολία. Κάτι άλλο τώρα. Εμείς απέσχουν από την ε, ψηφοφορία των ε, προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Συνεργασίας. Είπαμε ότι θεωρούμε ε, θετική την κατεύθυνση της ε, υπηρεσίας πνευματικής ιδιοκτησίας, ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, σύγκληση όσον αφορά την ε, αγορά, τη συνεργασία της κεντρικής υπηρεσίας αλλά και των γραφείων σε κάθε κράτος μέλος. Όμως είπαμε ότι οι δημοσιονομικές συνέπειες για αυτά τα προγράμματα ή έργα και η σχετική ενημέρωση δεν ήταν πλήρης. Άρα και εμείς δεν μπορούσαμε να έχουμε διαμορφώσει κάποια ε, πλήρη γνώμη. Οπότε και η διοίκηση είπε ότι πρόκειται να παρουσιάσει στη συνεδρίαση του Νοεμβρίου τα σχετικά στοιχεία. Όμως έγινε ψηφοφορία και σε εκείνη την ψηφοφορία εμείς οι δύο αποφασίσαμε να απόσχουμε. Η επόμενη συνάντηση τώρα θα γίνει στο Αλικάντε. Θα γίνει τον Νοέμβριο, 15 με 17 του μηνός. Η μέρη πρόκειται να παραστεί σε εκείνη την συνάντηση. Και μόλις έχουμε περισσότερη ενημέρωση για αυτήν την συνεδρίαση θα ενημερώσουμε την Επιτροπή μας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κυρία Χανίμπολ. Δεν έχω να ε, προσθέσω και τίποτα σε αυτά. Όμως, να λάβουμε υπόψη ότι εμείς ε, για αυτές τις δύο ψηφοφορίες ε, έχουμε απόσχη. Και Νομίζω ότι ο ρόλος μας ήταν επικοδομητικός. Θα πρέπει να προσέξουμε ακριβώς πώς έχουν οι εξελίξεις. Γιατί υπάρχουν εξελίξεις σε κάποια μέτωπα και σε άλλα δεν υπάρχουν. Και μας προβληματίζει αυτό. Θα προσπαθήσω να παραστώ στην επόμενη συνεδρίαση και να σας αναφέρω σχετικά. Γιατί αν συνεχιστούν αυτές οι εξελίξεις τότε θα πρέπει και εμείς να κάτσουμε και να προβληματιστούμε ακόμη περισσότερο πάνω σε αυτά. Ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρος. Υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις από τους ε, βουλευτές. Όχι, δεν ζητεί κανεί το λόγο. Επομένω, συνεχίζουμε και πάμε στο σημείο υπαριθμών 6. Ανταλλαγή απόψεων. Αυτό αφορά ε, στην ε, υιοθέτηση, θέσπιση ενός εργαλείου, ενός νομοθετήματος, το οποίο πρόκειται να συμβάλλει σε σταθερότητα και ειρήνη και εισηγητής ο κύριος Καβαντά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα αρχίσω με τα δύσκολα, αλλά είναι σημαντικό αυτό το ζήτημα. Περί τίνος πρόκειται. Θα πρέπει να κάνουμε μια επιλογή πια, παραδείγματο χάρη, αν η νομική βάση για μια πρόταση κανονισμού για ένα εργαλείο για τη συμβολή στη σταθερότητα και την ειρήνη είναι ναι ή όχι αποδεκτή ή πρέπει να τροποποιηθεί. Αυτό το μέσο, περίεργο ε, ε, αποτελείται από διάφορα μέτρα τεχνικής και οικονομικής ε, αρρωγής. Πρόκειται για την ε, συμβολή στην σταθερότητα και στην ειρήνη σε τρίτες χώρες και πρόκειται για όλους τους τομείς ε, της άμυνας ε, και ε, ακόμη και για το στρατιωτικό τομέα. Ο στόχος είναι η προστασία των ομάχων στις εμπόλεμες ζώνες, εκεί όπου υπάρχει κρίση, σε ευπαθείς περιοχές, για να ενθαρρύνουμε την οικονομική μεγέθυνση, την κοινωνική και ανάπτυξη, ανάπτυξη των περιβαλλοντικών μέτρων των αναπτυσσόμενων χωρών. Η νομική βάση που προκρίνεται για αυτή την πρόταση κανονισμού αποτελείται από την πρώτη παράγραφο του άρθρου 209 της ε, Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, από την παράγραφο 2 του άρθρου 212 επίσης, και αυτά τα δύο άρθρα είναι στο κεφάλαιο 3 που σχετίζεται με την συνεργασία με τις τρίτες χώρες και με την ανθρωπιστική βοήθεια. Ποιο είναι το ουσιαστικό πρόβλημα που τίθεται. Ένας τέτοιος ε, κανονισμός όμω θα έπρεπε να έχει ως νομική βάση μια διάταξη που σχετίζεται με την ε, κοινή ασφάλεια και την πολιτική άμυνα στις Ευρωπαϊκές Ένωσης ε, από ότι μια διάταξη που σχετίζεται με την ανάπτυξη, την αναπτυξιακή βοήθεια για την τεχνική και οικονομική βοήθεια. Έχοντας εξετάσει το θέμα, θα ήθελα να αρχίσω τη συζήτηση καταθέτοντας μία πρόταση. Εμείς ε, υπερασπιζόμαστε τη διατήρηση της ε, ισχύουσας νομικής βάσης για τους ε, λόγους που θα παραθέσω τώρα. Πρώτα απ' όλα, για τις συνθήκες έλλειψης σταθερότητας, για τις συγκρούσεις, ε, ελοχεύει ο κίνδυνος να πω σταθεροποιηθούν οι χώρες με τις οποίες έχει και διατηρεί εταιρικέ σχέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι Προφανές ότι είναι άρεκτη η σχέση ανάμεσα στην ασφάλεια και σταθερότητα σε μια χώρα και την ανάπτυξη αυτής της χώρας καθώς και την αναπτυξιακή βοήθεια. Από την εμπειρία μας βλέπουμε ότι τα μέτρα που συμβάλλουν στη διατήρηση ειρήνης και της σταθερότητας μπορούν να εκλειθούν ως μέτρα που συμβάλλουν επίσης στην ανάπτυξη, τον εκδημοκρατισμό και την ενίσχυση του κράτους δικαίου στις χώρες με τις οποίες έχει εταιρική σχέση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προβλέπει η πρόταση κανονισμού ότι αυτού του είδους η βοήθεια θα πρέπει να θεωρηθεί ως ίστατη λύση σε περίπτωση σοβαρής απειλής προς τα θεσμικά όρων, θεσμικού θεσμικούς φορείς μιας χώρας για την προάσπιση των θεμελιωδών ελευθεριών και των ε, βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν είναι τόσο αποδυναμωμένα αυτά τα κράτη σε μέτρο που δεν μπορούν να εγγυηθούν ε, αυτές οι βασικές ελευθερίες. Αυτό το μέσο θα το χρησιμοποιούμε για την ε, χρηματοδότηση, για την ε, στρατιωτική εκπαίδευση, για την ε, χρηματοδότηση που σχετίζεται με αγορά όπλων και πυρομαχικών. Από νομικής πλευράς, ο στόχος δεν είναι επιχειρησιακή βοήθεια προς στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά πρόκειται για τον τομέα της βοήθειας προς τις χώρες. Ε, θα έπρεπε ίσως να υπενθυμίσω ταυτόχρονα πως επιλέγοντας αυτή τη νομική βάση που σχετίζεται με την αναπτυξιακή βοήθεια και την τεχνική και οικονομική βοήθεια, εντασσόμεθα στη συνήθη νομοθετική διαδικασία ε, όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων και θα ήταν παράδοξο το Κοινοβούλιο να αποκλειστεί ε, από την εξέταση αυτής της νομικής βάσης. Ε, υπάρχει σχέση με την ε, κοινή πολιτική άμυνας ε, και ασφάλειας και εκεί ισχύει η ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου, διαφορετική δηλαδή διαδικασία και μεταβίας θα διαβουλεύονταν το Κοινοβούλιο και ενώ στην ουσία ότι θα γινόταν, θα ήταν δευτερεύουν ο ρόλος του Κοινοβουλίου και ετεροχρονισμένα θα γινόταν αυτή η διαβούλευση χωρίς καμία ε, σημασία. Με την συνήθεια όμως νομοθετική διαδικασία οι βουλευτές θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν ότι χρησιμοποιείται αυτό το μέσο για ανθρωπιστικούς λόγους ε, βάσει της κωδικοποίησης των πρακτικών που υποστηρίζει το Κοινοβούλιο κατά παράδοση. Προτού τοποθετηθείτε, θα ήθελα να ακούσουμε και τη νομική υπηρεσία που θα παραθέσει την επιχειρηματολογία, την επιχειρηματολογία της υπέρ της τροποποίησης νομικής βάσης και στη συνέχεια, Πρόεδρε, αν επιτρέπετε, θα ήθελα να ακούσω τη, τους συναδέλφους. Θα ήθελα να τοποθετηθούν έχοντας ακούσει και τη νομική υπηρεσία. Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Προτού δώσω το λόγο ε, στους βουλευτές, θα ήθελα να ακούσουμε τη νομική υπηρεσία. Παρακαλώ. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε δύσκολη υπόθεση, πράγματι κατανοούμε καλά τις ανησυχίες που εξηγεί ο εισηγητής και συμφωνούμε με την περιγραφή της καταστάσεως. Έχουμε βέβαια κάποιες αμφιβολίες σχετικά με αυτή τη νομική βάση. Για τον λόγο ότι το καθοριστικό στοιχείο για την επιλογή της νομικής βάσεως είναι οι συνιστώσεις, τα, συνιστώσα, τα συνιστώντα στοιχεία της νομικής πράξης. Πράγματι, η πολιτική αναπτύξεως φαίνεται να απαιτεί και κάποιο στοιχείο ασφαλείας. Αναγνώρισε και το δικαστήριο ότι μπορούν να ληφθούν μέτρα για την ασφάλεια στο πλαίσιο της αναπτυξιακής βοήθειας. Όμως, Εξετάζοντας τον στόχο εδώ της προτάσεως, σημειώστε ότι είναι και τροποποιητικό νομοθέτημα υφισταμένου κανονισμού, τροποποίηση στην οποία προβαίνει με την προσθήκη ορισμένων εξειδικευμένων στοιχείων. Όπως λέει λοιπόν ο εισηγητής, ο επικυρίαρχος στόχος είναι να επιτευθεί η βιώσιμη ανάπτυξη πιο συγκεκριμένος στόχος όμως εξακολουθεί να είναι ή υπό εξαιρετικές περιστάσεις και βεβαίως υπό τους περιορισμούς που εξήγησε ο να υπάρχει και ικανότητα, στρατιωτική ικανότητα σε τρίτες χώρες. Οι δε προβλέψεις που γίνονται αφορούν αποκλειστικά την δημιουργία στρατιωτικής ικανότητας. Να μην λησμονηθεί επίση ότι η δράση στο πεδίο τη εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλεία έχει ω στόχο την ασφάλεια. Στρατιωτικέ δράσει σε ευαίσθητε περιοχέ. Η αναπτυξιακή πολιτική, όπως και η τεχνική βοήθεια που προβλέπεται στο άρθρο 212, μπορούν να προσφέρουν τη νομική βάση, εάν δεν υπάρχει άλλη νομική βάση. Στο συγκεκριμένο τομέα εν προκειμένου, εμείς συμπεραίνουμε πάντως ότι το κέντρο βάρους εδώ είναι μάλλον η στρατιωτική πτυχή της ασφάλειας. Γι' αυτό σημειώνουμε αυτό ως προειδοποίηση, παρόλο που κατανοούμε ότι το Κοινοβούλιο επιθυμεί να κινηθεί μέσα στα πλαίσια της συνήθους, της τακτικής δηλαδή νομοθετικής διαδικασίας. Να υπενθυμίζω εν τέλει ότι έχουμε και το άρθρο 40 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ενώσεως που απαγορεύει πολιτικές της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας να επηρεάζουν πολιτικές της Ένωσης. Αλλά και το αντίθετο. Πολιτικές της Ενώσεως επηρεάζουν πολιτικές πά. Άρα εδώ μπορεί να οδηγηθούμε σε δυσκολίες. Βέβαια, εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά από το προηγούμενο άρθρο, το 47 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο κρατούσε την κοινή εξωτερική πολιτική εκτός κοινοτικών πολιτικών. Τώρα όμως είναι αμοιβαία εξαρτώμενες. Άρα εδώ πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Για αυτό το λόγο διαπιστώνουμε εμείς ότι υπάρχει ενδεχομένως ένα πρόβλημα με την επιλογή αυτής της νομικής βάσης. Ένα σημαντικό σχόλιο ακόμη, τελευταίο, είναι εμείς αξιολογήσαμε την πρόταση ως έχει. Πριν να συζητηθεί στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Ίσως υπάρχουν και άλλες προθέσεις σχετικά με, την, με το περιεχόμενο της προτάσεως. Αλλά πάντως, ε, εν ολίγης θεωρούμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την προτινόμενη νομική βάση. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Κύριε Χαούταλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σημαντικό θέμα και σημαντική χρονική στιγμή, διότι για πρώτη φορά νομίζω ακούμε την νομική υπηρεσία ενός θεσμικού οργάνου να μιλεί δημοσία και να εκφράζει επιφυλάξεις αλλά και απόρριψη της επιλογής νομικής βάσης για τη συγκεκριμένη τροποποίηση του κανονισμού την οποία παρουσίασε στις 15 Εβδόμου η πάτη εκπρόσωπος Μογκερίνη. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι και όπισθεν και κρυσμένων θυρών και οι νομικέ υπηρεσίε των δύο άλλων θεσμικών οργανών έχουν εκφράσει τι ίδιε επιφυλάξει. Και βεβαίω αυτά πρέπει να τα βλάβουμε σοβαρά υπόψη. Και εγώ κατανοώ ότι υφίστανται αυτέ οι ανησυχίε, δηλαδή ότι πρέπει κάτι τι να κάνουμε ώστε να υποστηρίξουμε αυτές τις ευάλωτες χώρες για να αντιμετωπίσουν καταστάσεις συγκρούσεων, να μην καταρρεύσουν, να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των πληθυσμών τους. Όμως, όπως είπε και η νομική υπηρεσία, ο παρόν μηχανισμός αφορά κυρίως την προσθήκη ενός στοιχείου που αφορά καθαρά τη στρατιωτική υποστήριξη με εξαίρεση όπλων και πυρομαχικών. Βέβαια, μπορεί ωστόσο να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία στρατιωτικών βάσεων από τη σκοπιά της αναπτυξιακής βοήθειας που και από τη δική μου εμπειρία αναδεικνύεται πολύ σημαντική, πρέπει να αναρωτηθούμε αυτό πραγματικά χρειάζεται να κάνουμε. Δηλαδή σε αυτά να δαπανίσουμε τους πόρους της Ένωσης που προβλέπονται για την αναπτυξιακή βοήθεια. Η απάντηση που δίνω εγώ είναι όχι. Κατανοώ τον πειρασμό που αντιμετωπίζει το Κοινοβούλιο για την διατήρηση δηλαδή των προνομίων του, αλλά να αντισταθούμε στον πειρασμό αυτό. Ακόμα και αν αυτό αποβεί σε βάρος της δικής μας ας πούμε άνεσης, διότι πρόκειται στην ουσία για μια απόπειρα να περιβληθεί και πάλι τον διακυβερνητικό μανδύα η συνεργασία αυτή. Το ιστορικό της προτάσεως δείχνει ότι η πίεση προς την κατεύθυνση αυτή αρχίζει το 2011 και, και μάλιστα έχει ξεπεράσει κάθε όριο από τότε με ένα, μια κέρια στιγμή μια επιστολή στις 15 Τετάρτου από ένα αριθμό χωρών μελών που απευθύνθηκε στην ύπατη εκπρόσωπο να τροποποιήσει ταχύτατα την πρόταση, τον κανονισμό δηλαδή, συμβολής σε ειρήνη και σταθερότητα προς την κατεύθυνση αυτή. Νομίζω θα είναι κρίμα να, να ακολουθήσουμε μοναχά τη λογική των προνομίων του Κοινοβουλίου, να δείξουμε το θάρρος να εξετάσουμε περισσότερο σε βάθος το θέμα αυτό. Άλλωστε ξαναλέω, οι νομικές υπηρεσίες και των τριών θεσμικών οργάνων στέκονται πολύ επικριτικά και με επιφύλαξη απέναντι στην πρόταση αυτή. Και μόνο αυτή τη στιγμή η Μογκερίνη έβαλε τον επικεφαλής του προσωπικού του γραφείου να ασχοληθεί, πήγε και η υπόθεση αυτή στο ΔΕΦΚΟ, δηλαδή στο Τμήμα Αναπτυξιακής Βοήθειας. Ας έχουμε λοιπόν υπόψη και το ενδεχόμενο να απορρίψει η Επιτροπή μας την προτινόμενη νομική βάση. Ο κ. Βος. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κατανοώ τα επιχειρήματα της κυρίας Χάουταλα όπως και της νομικής υπηρεσίας. Όμως από την άλλη μεριά οφείλω να διερωτηθώ μήπως έχουν αλλάξει οι καιροί. Ασφαλώς βρισκόμαστε στα όρια από νομική σκοπιά. Μήπως όμως έχει έρθει η ώρα ε, να κάνουμε και κάτι διαφορετικό και να ακολουθήσουμε μια ρεαλιστική προσέγγιση. Διαρωτώ με, εάν δεν τα πράξουμε αυτά που λέμε εδώ, μπορούμε καν να προσφέρουμε αναπτυξιακή βοήθεια σε χώρες οι οποίες έχουν γίνει σχετικά ασταθείς, δηλαδή θα παρακολουθούμε απλώς χώρες τις οποίες προσπαθούμε να σταθεροποιήσουμε μέσω της αναπτυξιακής βοήθειας, απλά να γίνονται ασταθείς. Γι' αυτό και θεωρώ ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα αυτό περισσότερο. Μήπως δηλαδή τα παρακολουθήματα ή μέσα στα πλαίσια ας πούμε, των παρακολουθημάτων της αναπτυξιακής βοήθειας πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας και εδώ, αλλά στα συγκεκριμένα καθήκοντα. Δεν βλέπω να υπάρχει άλλη δυνατότητα επιλογής. Βλέπουμε ανά τον κόσμο πολλές ασταθείς χώρες, περιφέρειες, όπου θα έπρεπε να πούμε και για το δικό μας καθαρά συμφέρον ότι πρέπει να τις βοηθήσουμε να σταθεροποιηθούν. Να υπάρχει όμως η δυνατότητα να συνοδεύονται και να διασφαλίζονται τα μέτρα αυτά αναπτυξιακής βοηθείας και με τις ενέργειες που συζητούμε. Αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες. Νομικά θεωρώ ότι μπορεί να ερμηνευθεί με τον τρόπο αυτό. Σύμφωνοι είναι κάπως εωριακό. Αλλά επαναλαμβάνω ότι σήμερα πλέον οι καταστάσεις είναι διαφορετικές από ό,τι ήταν κάποτε όταν είχαν δημιουργηθεί αυτές εδώ οι νομικές βάσεις. Χρειάζεται λοιπόν να εξελίξουμε κι εμείς τον τρόπο αντιμετώπισης και ίσως η προτινόμενη ε, δυνατότητα να είναι η ορθή. Εάν μπορούμε δηλαδή να διατηρήσουμε τον στόχο, θα πρέπει αυτό να μπορεί να γίνει και μέσα σε αυτούς τους αβέβαιους καιρούς. Και γι' αυτό εν τέλει θεωρώ την προσέγγιση Καβαδά ορθή. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Παρακολούθησα προσεκτικά τα εκατέρωθεν επιχειρήματα και ομολογώ ότι τελώ εν Συζητούμε δηλαδή για τη νομική βάση. Άρα κανονικά η σύντηση αυτή είναι νομικού χαρακτήρα. Δηλαδή στρέφεται γύρω από το ερώτημα ποια είναι η σωστή νομική βάση. Οι εξηγήσει της νομικής υπηρεσίας δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρες. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να μας δώσουν μια τοποθέτησή τους γραπτή, ίσως και από άλλες νομικές υπηρεσίες, ώστε να έχουμε μια ιδέα. Και πάνω σε αυτό έρχεται και μια συζήτηση τώρα για τα προνόμια του Κοινοβουλίου, που και αυτό αποτελεί πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, και υπάρχει και μια συζήτηση πλέον για τα μέσα, τους μηχανισμούς της αναπτυξιακής βοήθειας. Βρίσκω ότι είναι πλήθος των στοιχείων αυτών και δεν θα πρέπει να καταχραστούμε τα νομικά επιχειρήματα για να υπερασπιστούμε την α ή τη β θέση. Είναι χρήσιμο λοιπόν, επαναλαμβάνω, να έχουμε γραπτό στην τοποθέτηση της νομικής υπηρεσίας, ώστε να τη μελετήσουμε πριν να μπορέσουμε να κάνουμε τα επόμενα βήματα στη διαδικασία αυτή. Ευχαριστώ κύριε ε, Πρόεδρε. Η κυρία Τελβό επειδή συνήθω δεν ασχολούμαι με, με νομικές βάσεις, γιατί εγώ ασχολούμαι με την ε, ε, γονική άδεια. Δεν γνώριζα ότι υπάρχει υπάρχει ε, η τοποθέτηση τη νομική υπηρεσιας υπηρεσίας από 31η 8. Ε, ζητώ συγγνώμη γιατί δεν έχω διαβάσει. Αλλά ε, θεωρηθούν τα λόγια μου σαν τοποθέτηση που λέει ότι χρειαζόμαστε ακόμα κάποιο χρόνο μέχρι ότου κατασταλάξουμε. Ο κύριος Καβαδά, Καβαδά. Ευχαριστώ αγαπητέ πρόεδρε. Χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα υπήρχε σήμερα πλέον Παλαιστινιακή Αρχή. Θα υπήρχε ένας αριθμός προσώπων χωρίς καμία διοικητική βάση. Διεξήχθησαν στρατιωτικές επιχειρήσεις σε διάφορα σημεία του περιβάλλοντος χώρου μας, ιδίω στη Μεσόγειο, όπου είδαμε καθαρά τα όρια τους. Και Είμαι γνώμη στον κύριο Βος που εξήγησε πόσο πολύ έχει αλλάξει σήμερα η γεωπολιτική κατάσταση. Δεν είναι θέμα πλέον να δούμε εάν ναι ή όχι το κοινοβούλιο θα πρέπει να ακουστεί, να είναι συμβουλευτική ή όχι γνώμη του κτλ. Η νομική υπηρεσία καλείται να ενισχύσει τη θέση μας, να μας διαβεβαιώσει ότι θα δημιουργήσει μία νομική βάση που θα μας επιτρέψει να αναλάβουμε πλήρως τον ρόλο μας ως ε, εκλεγμένοι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών λαών απέναντι στην διοίκηση, στην ευρωπαϊκή διοίκηση. Και σε αυτούς τους δύο καιρούς όπου από κάποιες απόψεις υπενθυμίζει και το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1930 είδαμε πολλούς να λένε ότι το νομικό πλαίσιο δεν επιτρέπει το ένα ή το άλλο, όπως και τότε. Αυτοί που ε, επιζητούν την ειρήνη και με στρατιωτικά μέσα πρέπει να επιτρέψουν την εξασφάλιση της ειρήνης και με άλλα μέσα. Εάν δεν υπάρχει βοήθεια και αν δεν υπάρχουν δομές από πίσω, οποιαδήποτε στρατιωτική βοήθεια δεν αρκεί. και καταλήγουμε στο χάος. Αυτό είναι το ερώτημα που τίθεται εν τέλει. Πρώτο λοιπόν. Θα ασχοληθούμε με το μέλλον της Υπήρου μας, με επιχειρήσεις που είναι εκτός των ορίων μας και θα ασχοληθούμε με την ανθρωπιστική βοήθεια όταν θα είναι αναγκαίο. Και υπάρχει και μια δεύτερη ερώτηση που οφείλουμε να θέσουμε. Η εξή. Είναι νοητό όπως είναι τα πράγματα σήμερα με τους ε, λαούς της Ευρώπης να δεχθούν να γίνει μια στρατιωτική επιχείρηση χωρίς ξεκάθαρη ψήφο του Κοινοβουλίου. Για μένα αυτό είναι αδιανόητο. Η απάντησή μου είναι λοιπόν αρκτική. Υπό την έννοια αυτή θέλω να κάνω την εξή πρόταση στην ε, νομική υπηρεσία. Και αναμένω βεβαίως να ακούσω και τις απόψεις όλων των συναδέλφων. Διότι στόχος είναι να συντάξουμε έκθεση η οποία να απηχεί όλες τις απόψεις απέναντι στην διοίκηση. Δηλαδή, εάν θα υπάρξει στρατιωτική ή όχι παρέμβαση, διότι ο ρόλος μας είναι αυτός. Η στήριξη των κρατών. Θα έχω λοιπόν να κάνω την εξή πρόταση. Ή θα μας δώσετε μία νομική βάση, αλλά νομική υπηρεσία, που θα επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε, να διαχειριστούμε τα νέα αυτά προβλήματα. Θα φροντίσετε όμως να διασφαλίσετε ότι το Κοινοβούλιο θα μπορεί να τοποθετηθεί, να εκφραστεί και να ψηφίσει. Ή κάτι τέτοιο σας είναι αδυνάτον, οπότε εγώ προτιμώ να μην αλλάξω άποψη. Διότι ό,τι έχουμε, έχουμε. Κρατούμε στα χέρια σας. Θα ακούσουμε λοιπόν την πρότασή σας και θα δούμε τι μπορεί να προσφέρει. Αυτό ήθελα να απαντήσω λοιπόν και στους συναδέλφους και στην νομική υπηρεσία. Η νομική υπηρεσία θα πρέπει να μας βάλει τις ράγες για να, μπορέσουν, για να μπορέσει ο προβληματισμός μας να προχωρήσει. Ο πρόεδρος, η νομική υπηρεσία. Θα είμαι σύντομος. Αυτά που εξήγησε ο εισηγητής αντιστοιχούν στις δικές μας απόψεις. Δεν είναι τα πράγματα ως συνήθως. Η εξωτερική πολιτική είναι άλλο θέμα. Άρα ε, εκεί δεν έχουμε αρμοδιότητα, αλλά έχω να σας πω μόνο το εξή. Για να είμαστε δημιουργικοί πρέπει να σας πούμε ότι εμείς αξιολογούμε αυτή τη ε, διαδικασία ως έχει και ακριβώς εκεί είναι και το πρόβλημα. Δεν μπορώ να αλλάξω την ανάλυση, γιατί αυτή μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχουν και άλλες αναλύσεις που μπορεί να κάνει κάποιο άλλος, αλλά εμείς αυτή την ανάλυση κάνουμε. Τώρα όσον αφορά το τι γίνεται στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, ίσως το περιεχόμενο αυτού του ε, νομοθετήματος θα μπορούσε να τροποποιηθεί και θα μπορούσε να εξελιχθεί ούτως ώστε να προσαρμοστεί με την πολιτική Ανάπτυξη. Οπότε τώρα δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στις λεπτομέρειες, γι' αυτό είναι δική σας δουλειά. Μετά όμως να κάνουμε άλλη μια αξιολόγηση. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα. Απλώς να προβληματιστούμε πάνω σε αυτό. Να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν. Uh, Mrs. Yeah, thank you very much. Uh, Κύριε Χάουταλα, ευχαριστώ πολύ. Μου φαίνεται ότι όλα αυτά συζητούνται στην Επιτροπή Ανάπτυξη και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Όμω, εμεί εδώ συζητούμε τη νομική βάση, τι προβλέπεται από τι ε, συνθήκε. Οπότε θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε το ότι ε, η κάθε επιτροπή αλλιώ θα δει το θέμα. Νομίζω όμως ότι η κυρία Ντελβό έχει δίκιο. Τώρα χρησιμοποιείται έτσι η νομική βάση, ούτω ώστε αυτό να καταλήξει σε κάτι χρήσιμο. Και οπωσδήποτε υπάρχει σχέση εδώ με την πολιτική εξωτερικών, με την πολιτική εξωτερικών σχέσεων, γιατί και στη χώρα μου είχαμε ε, φιλοξενήσει μια σημαντική διάσκεψη που αφορούσε ε, την ανάπτυξη και είχε σχέση με αυτό. Δηλαδή υπάρχει αυτή η σχέση ασφάλειας και ανάπτυξης, οπότε πώς να αλλάξει κανείς άρδιν αυτή τη σχέση την ε, Αναπτυσιακή συνεργασία, δηλαδή το ώστε να αντιμετωπιστεί η φτώχεια, να δημιουργηθούν κάποια άλλα προβλήματα όπως η αλλαγή του κλίματος, ε, η έλλειψη παιδείας για τόσους πολλούς ανθρώπους, ε, άλλα θεσμικά ζητήματα, γιατί θα μπορούσε κανείς να μετελθεί και άλλα μέσα συμμετοχή σε στρατιωτικέ επιχειρήσεις κλπ. Όλα αυτά επιδέχονται συντονισμό και υπάρχει μια ε, σφαιρική γενική στρατηγική τη Ένωση και εκεί θέλουμε να υπάρξει συντονισμός. Όμως, δυστυχώς, η λόγω πρόταση, δυστυχώς λέγω προσπαθεί να ε, χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο συνεργασίας και ανάπτυξης για μια συγκεκριμένη χρήση. Δηλαδή, αυτά τα 100 εκατομμύρια είναι πολλά λεφτά. Όμως, ποιος ξέρει εάν θα βρεθούν και άλλα χρήματα για τον τίτλο 4. Γιατί ίσως κανείς θελήσει να πάρει και άλλα χρήματα από τον προϋπολογισμό της αντισιακής πολιτικής. Αλλά να μην ξεχνούμε τι προβλέπει η συνθήκη για αναπτυξιακή βοήθεια και συνεργασία. Να μην ξεχνούμε και τι αρμοδιότητε του Κοινοβουλίου, γιατί το πρωτογενέ κοινοτικό δίκαιο δεν μπορούμε να το αλλάξουμε και αν λέμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει περισσότερε αρμοδιότητε όσον αφορά ε, την ε, ΚΕΠΑ ή την Επιτροπή Ανάπτυξη. Βεβαίω και θέλουμε περισσότερη συμμετοχή ε, για την κοινή ε, επιτροπή, για την κοινή πολιτική ε, εξωτερικών σχέσεων κλπ. Όμως τώρα δεν μπορούμε αυτό να το κάνουμε με την τροποποίηση της νομοθεσίας για αυτά τα εργαλεία. Ο εισηγητής πρότεινε κάτι πολύ αξιόλογο να δούμε τις γνωμοδοτήσεις των νομικών υπηρεσιών Συμβουλίου και Επιτροπής. Πολύ σημαντικό. Επίσης ε, και οι πολίτες θα πρέπει να ξέρουν τι γίνεται. Οπότε θα πρέπει για πρώτη φορά αυτά που μας απασχολούν ε, εδώ στην Επιτροπή μας να είναι ε, κάτι που να το, να το μάθει ο κόσμος, ο πρόεδρος. Να ψηφίσουμε όσον αφορά τη σχετική πρόταση όμως θα μπορούσαμε να αναβάλουμε την ψηφορία για την επόμενη συνεδρίαση, αν δεν έχετε αντίρρηση, ούτως ώστε όλοι να μπορούν μέχρι τότε να έχουν διαμορφώσει μία άποψη για αυτό το σημαντικό ζήτημα. Οπότε αναβάλουμε την ψηφορία για την επόμενη συνεδρίαση. Uh, now, uh, the next items 7, 8 and... 7, 8 και 9. Τα επόμενα θέματα τα οποία όμως αναβάλλονται. Πάντως, σας ενημερώνω ότι η προθεσμία για τροπολογίες είναι η 8η Σεπτεμβρίου μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και τώρα. Συνεχίζουμε με το θέμα υπαριθμών 10. Δηλαδή θα γίνει η συζήτηση ενό και δύο εκθέσεω όσον αφορά τι ε, δηλώσει οικονομικών συμφερόντων των ε, επιτρόπων. Τον λόγο έχει τώρα ο κύριο Μπυρόν που είναι ο εισηγητή. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να μην μακρηγορήσω. Για που έχουμε τόσο να συζητήσουμε αυτό το θέμα θα έπρεπε να μας ε, βοηθήσει να καταλήξουμε σε κάποια τοποθέτηση συνενετική και αρκετά μετριοπαθή. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί επανειλημμένα έχει διατυπωθεί από πλευράς μου κάποιος φόβος. Και δεν θέλω, λέω ο παγίος να γίνει η Επιτροπή μας δικαστήριο. Άρα δεν θέλουμε να αλλάξουμε το ρόλο του Κοινοβουλίου ή της Επιτροπής μας. Άρα να μην καταλήξουμε σε κάτι μαύρο ή άσπρο για αυτό το θέμα. Απλώς να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε κάτι. Κάτι επί του οποίου πρόσφατα είπαμε ότι η κατάσταση δεν είναι και τόσο ικανοποιητική. Λέω ότι δεν θέλουμε να το αλλάξουμε, δεν θέλουμε βάθρων να τα ανατρέψουμε ό,τι προβλέπεται, απλώς να βελτιώσουμε. Οπότε και εν προκειμένου νομίζω ότι υπάρχει μια συνένεση και η καθημερινή βασική γραμμή που ήταν και η δική μου είναι ότι το Κοινοβούλιο να μπορέσει να ασκήσει τις αρμοδιαιτές του πλήρως στα πλαίσια της θεσμικής ε, ισορροπίας. Οπότε και εμείς να μπορέσουμε να κινηθούμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας αλλά και να τις ασκήσουμε πλήρως ώστε να γίνει σεβαστό το κοινοβούλιο και αρμοδιοτήτες του. Και είπαμε ότι στα πλαίσια αυτά η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων να μπορέσει και αυτή να επιτελέσει το ρόλο που της έχει ανατεθεί. Οπότε και έτσι το Κοινοβούλιο μας έχει αναθέσει κάτι το συγκεκριμένο. Και θα πρέπει έτσι και εμείς να ενεργήσουμε και να είμαστε αποτελεσματικοί. Είπαμε, ο ρόλος μας δεν είναι να γίνουμε δικαστήριο, ούτε να κάνουμε κάποιο είδους ε, έρευνες και ανακρίσεις. Απλώς θα πρέπει να ε, επιλύονται τα ζητήματα σύγκρουσης οικονομικών συμφερόντων εν προκειμένου για τους επιτρόπους. Οπότε υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι ειδικοί, οι οποίοι δεν πρέπει να μένουν έξω από αυτό το έργο. Η σύγκρουση μόνο δεν είναι σύγκρουση αρμοδιοτήτων. μπορούσε επομένω ε, σε κάθε περίπτωση να έχουμε να κάνουμε με κάποιον άριστο επίτροπο. Θα πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι περιχαρακώνεται πάρα πολύ καλά τι είναι η σύγκρουση οικονομικών συμφερόντων και θα πρέπει να φροντίσουμε εμείς ούτως ώστε να μην υπάρχει κάποια σκιά που δυσκολεύει το έργο κάποιου επιτρόπου και σε αυτό επιμένω αυτό, αυτό θα πρέπει να κάνουμε επ' αυτού θα πρέπει να έχουμε την έκθεση που να είναι συνετική. γι' αυτό με απασχολεί Επομένω, δεν θέλω τώρα να επισέλθω στις λεπτομέρειε, γιατί έχουμε και άλλα θέματα σήμερα να συζητήσουμε σήμερα Απλώ θα ήθελα να ε, μπορέσουμε, επί τη βάση της εκθέσεώς μου, η εξέταση τη σύγκρουση συμφερόντων να μελετηθεί με τέτοιον τρόπο μέσα σε αυτή την ε, συγκυρία όπου του πολλές επικρίσεις κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην οδηγηθούμε σε αντιπαράθεση του γενικού συμφέροντος με το προσωπικό. Και να δούμε το πώς θα μελετήσουμε ακριβώς ε, το θέμα υπό το φως της διάκρισης του γενικού συμφέροντος από το συγκεκριμένο ή το προσωπικό. Και λέμε τώρα για το ότι έχουν διατυπωθεί κάποιες ε, επιφυλάξεις και για την πολιτικοποίηση του θέματος αλλά όχι η έκθεσή μου ε, δεν είναι ένα κείμενο ε, φορτισμένο πολιτικά απλώς λέω ότι θα πρέπει τη δουλειά μας να την ε, διέπει η διοντολογία και προκειμένου όπως και γενικότερα άρα θα πρέπει να βελτιώσουμε τις σχετικές δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων αυτές που κατατίθενται στην αρχή της ε, θητείας όσον αφορά τα οικονομικά σχέδια της οικογένειας ενός επιτρόπου και δεν αναλύουμε το τι τις αρμοδιότητες του επιτρόπου αυτό είναι θέμα αρμόδιας επιτροπής γιατί σας επαναλαμβάνω δεν θέλουμε να δικάσουμε κάποιον απλώς θέλουμε κάθε φορά να αντλούμε τις ε, δέουσες πληροφορίες επίσης ε, δεν επιβάλλουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνουμε, προτείνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βελτιώσει κάποια στοιχεία. Πρώτη φορά ασχολούμαι με αυτό για να μην έχουμε κάποιο είδου σύγκρουση μεταξύ της αρχικής δήλωσης του κάθε επιτρόπου και από την άλλη μεριά το τι γίνεται ε, κατά την άσκηση των συμφερόντων του όσον αφορά τα οικονομικά συμφέροντα της οικογένειας του. Με μεγάλη προσοχή περιμένουμε τις προτάσεις σας ούτως ώστε το κοινοβούλιο να μπορέσει να ασκήσει το ρόλο του σαν αφορά αυτέ τι αξιολογικές κρίσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, προσυπογράφω και την, και την τελευταία λέξη του εισηγητού. Είναι σωστή η κατεύθυνσή του. Κάθε άνθρωπος και βεβαίως και επίτροποι και υποψήφοι επίτροποι ε, ε, διαθέτουν ιδιωτικά συμφέροντα. Αλλιώ θα έπρεπε να βρούμε πράσινα ανθρωπάκια από τον Άρη για να του διορίζουμε επιτρόπου. Δεν πρόκειται γι' αυτό. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να αναλύσουμε πού βρίσκεται το πραγματικό ενδιαφέρον, το γενικό, το, το συνολικό συμφέρον και πού είναι τα ε, ιδιωτικά συμφέροντα. Λοιπόν, θεωρώ ότι αυτά που προτείνετε, αγαπητέ συγκητά, μπορώ να τα υποστηρίξω. Τώρα, έχω ορισμένα σχόλια σε, για συγκεκριμένους τομεί προβλημάτων. Το Κοινοβούλιο πρέπει με συνέστημα ευθύνης να προβεί στους ελέγχους εκτελών το καθήκον του και όχι τραλαλά, δηλαδή να αναλάβει επίσημο ρόλο. Όχι να δει τώρα εάν και η τελευταία δήλωση έχει ε, συμπληρωθεί σωστά, χωρίς να παίξει και τον ρόλο του δικαστού. Αλλά να μην ξεχάσουμε και τα μέλη οικογενειών, διότι έχουμε κάποιες εμπειρίες σχετικά. Έχουμε τις εμπειρίες από τα Lux Leaks, καθώς και από την Εξεταστική Επιτροπή για τα έγγραφα του Παναμά, όπου λάβαμε κάποιες πληροφορίες και γνωρίζουμε ότι σήμερα για πολλές επιχειρήσεις αλλά και για πολλά, πολλούς πλούσιους ιδιώτες είναι σύνηθες να βάζουν μέλη οικογενειών, των οικογενειών τους δηλαδή, να έχουν αυτά, δηλαδή στην κατοχή τους μετοχές ή κάτι άλλο, περιουσιακά στοιχεία ή εταιρείε κλπ. Ενώ στην πραγματικότητα να κρύβονται πίσω από τα πρόσωπα αυτά άλλα πρόσωπα. Μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων μας, της άσκησης των καθηκόντων μας, δηλαδή εξέτασης έρευνας, δεν θα παίξουμε τον ρόλο βέβαια του δικαστού, αλλά όχι να περιοριστούμε και μονάχα σε μια τυπική επιτήρηση, να δούμε δηλαδή αν όντως συμπληρώθηκαν σωστά οι δηλώσει, αλλά να το εξετάζουμε και επί τη ουσία. Όπω δηλαδή πρότεινε ο εισηγητή, βρίσκω ότι αυτά που είπε βαίνουν στην σωστή κατεύθυνση. Να προσέξουμε ιδιαίτερα τι διατυπώσει μα. ώστε να μην δημιουργήσουμε απλά ένα πλαίσιο και να αποφύγουμε να μπουν στην υπόθεση αυτή τα μέλη της οικογένειας μέχρι και του 17ου βαθμού και ξαφνικά να βάλουν αυτοί οι πονηροί επιχειρηματίες κάποιον φίλο τους να ε, παίξει τον άνθρωπο. Εσείς κύριε Καβάντα. Πρώτα απ' όλα θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Συμφωνώ πολύ με τις ε, διευκρινήσεις του κυρίου Ντυρά σε σχέση με το ρόλο του εγγράφου αυτού. Δηλαδή, να διευκρινίσουμε ότι θα πρέπει να γίνονται σεβαστές ε, κάποιες βασικές αξίες. Θα δούμε στη συνέχεια αν είναι δυνατόν ε, πλήρω να τον υποστηρίξουμε, ίσως τροποποιήσουμε κάποιες λεπτομέρειες, αλλά δεν θα έχω κανένα πρόβλημα να τον υποστηρίξω. Λοιπόν, τώρα πέρα από την εμπειρία, όπως είπαν και οι δύο συνάδελφοι, ο κύριος Τυράν και η κυρία Ρέγνερ, θα ήθελα να μην ε, εκτροχιαστούμε με τις αξίες αυτές, ε, ενώ απειλείται η Ευρώπη από αυτό το κίνημα του εθνικισμού. Θα ήθελα να παραπέμψω στον Επίτροπο Μποτιλιώνε, που μας είχε παρουσιάσει ο κύριος Μπερλουσκόνη, οι παλιοί θα το θυμούνται, μας τον είχε παρουσιάσει ως υποψήφιο επίτροπο για τις πολιτικές ελευθερίες, για να προεδρεύει για να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο στην Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή για ε, τα θέματα ΤΖΑΙ, δηλαδή δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις. Και ξεκάθαρα ε, αυτός ο διανοούμενος δρομέος ήταν ομοφιλόφοβος, ξεκάθαρα ξενόφοβος και ήταν σχεδόν κόλαφος που η Ιταλική κυβέρνηση ήθελε να μας κάνει να καταπιούμε αυτό το πικρό χάπι. Μετά από τους δύο ακροάσεις επέμεναν. Τέλος πάντων τότε, και το λέω αυτό διότι είναι πολύ παλιό αυτό το ζήτημα, μας απασχολεί εδώ καιρό. Ε, το λέω όμως διότι εμείς δεν έχουμε κανένα μέσο για να εξακριβώσουμε τις δηλώσεις. Δεν είμαστε δικαστήριο εδώ. Οπότε γινόμαστε συνένοχοι κατά παράληψη αυτών των ψεμάτων που δηλώνουν, ε, δηλώνονται ε, ενίοτε ενώπιον του Κοινοβουλίου. Οπότε θα πρέπει να διευρυνθούν διατάξεις ούτως ώστε ε, ακούσια να μην γινόμαστε συνένοχοι. Τρίτον. Έχω την εντύπωση πως είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι παρότι δεν είμαστε δικαστήριο, διαβιβάζουμε την ε, ειλικρίνεια. Δεν πρέπει λοιπόν να ε, περιπέσουμε σε ένα ε, παράλληλο σύμπαν ανηλικρίνειας. Και όπως είπε και ο Πρόεδρος νωρίτερα, όταν υπάρχει αυτός ο στρόβιλος υποψιών, παρασύρεται το Κοινοβούλιο σε αυτές τις ε, υποψίες λόγω της κακής οργάνωσης του ε, ρυθματολογίου. Και δεν υπάρχει αρκετή σαφήνεια για το ζήτημα, διότι ε, δεν οργανώνεται με αρκετή σαφήνεια η ακρόση ενώπιον της Επιτροπής μας. Και γι' αυτό θα συμφωνήσω και πάλι με τον κύριο Ντυρό, ενδεχομένω ε, να ε, συγγυθώ κάποια πρόσθετα στοιχεία, αν μου επιτρέπετε. Το θέμα της ειλικρίνειας, ε, ε, απόλυτης ειλικρίνειας σε σχέση με τις δηλώσεις που κατατίθεται ενώπιον του Κοινοβουλίου για να βγούμε από αυτόν τον κόσμο της υποψίας που πλήττει τη φήμη του Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε κύριο Ζεύκα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντιρό για την έκθεση που μας παρουσίασε. Είναι εξαιρετικά επίκαιρο το ζήτημα και είναι συναισθηματικά φορτισμένο το ζήτημα διότι μεταξύ άλλων υπάρχει και μία επιθυμία να, από κάποιους να κάνουν πολιτικά παιχνίδια Εκτιμώ αυτά που είπαν οι συναδέλφοι. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλά ενάψματα για τη συζήτηση και το μελλοντικό προβληματισμό μας, ούτως ώστε να καταλήξουμε σε μια απόφαση. Ε, στρέφουμε προς τον κύριο Καβαντά. Θα μπορούσατε να μου διευκρινίσετε ακριβώς σε ποιες περιπτώσεις το Κοινοβούλιο κατέστη συνένοχο σε οποιαδήποτε ψέματα, απάτες. Εγώ είμαι πολλά χρόνια στο Κοινοβούλιο και δεν θυμάμαι κάποια τέτοια περίπτωση. Θα ήθελα λοιπόν να μας μιλήσετε, να μας δώσετε συγκεκριμένα παραδείγματα για τέτοιες πράξεις. Δώσα το παράδειγμα του κυρίου Βοτιλιώνη. Να λοιπόν, είναι η αυτή απόδειξη του, της εξουσίας που έχει το Κοινοβούλιο. Ε, να μπορούσαμε να πούμε στην Ιταλική κυβέρνηση, ευχαριστούμε για τον διοριστέντα υποψήφιο, στείλτε μας όμως κάποιον άλλον γιατί δεν μας κάνει. Οπότε δεν πρόκειται σε κάποια μεμπτή πράξη. Το ίδιο συμβαίνει και με την δεύτερη επιτροπή του Μπαρόσο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν υπήρξε καμία έκνομη πράξη. Δεν Αλλού έγκυται το πρόβλημα και θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά που είπε ο εισηγητής, ο Πασκάλ Ντυρό. Συμφωνώ απολύτως με την ανάλυση του. Διαφωνώ όμως, Πασκάλ, με πάρα πολλά στοιχεία που σε περιέλαβες στην έκθεση, διότι δυστυχώς έτσι θα δοθεί μια πλημελής εντύπωση στους αναγνώσεις. Πολύ διαφορετική από αυτή που δημιουργείται στους ακροατές σημερινή συνεδρίαση με την παρουσίασή σου. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχουμε μια ευρεία θέσμη ε, εργαλείων για να εξακριβώνουμε την ακρίβεια των δηλώσεων ε, και των απαντήσεων σε αυτό το ρυθματολόγιο. Όμω ας μην γίνουμε, ας μην χειραγωγηθούμε σε αυτά τα πολιτικά παιχνίδια. Δεν είμαστε εξεταστική επιτροπή ούτε εισαγγελία θέλουμε να εξακριβώνουμε ε, την ε, ακρίβεια αυτών των εγγράφων που μας διαβάζετε βάσει του ιστορικού κανονισμού του Κοινοβουλίου και τη Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για να μπορέσει να διοριστεί κάποιος επίτροπος. Αυτό είναι ο στόχος μας. Δεν μπορούμε όμως ε, να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή το Κοινοβούλιο δεν θα φτιάξει καινούριο ερωτηματολόγιο που θα πρέπει να συμπληρώνουν οι, οι δόριες επίτροποι. Δεν είναι δική κόσμος ο ρόλος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να τροποποιήσει το ερωτηματολόγιο και πώς μπορούμε να την υποχρεώσουμε ζητώντα να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Να μην ε, λαμβάνουμε προφορές σε σχέση μόνο με τα οικονομικά συμφέροντα του ιδίου του υποψηφίου, αλλά και τη οικογένεια του. Εμεί δεν είμαστε σε θέση να τροποποιήσουμε το ερωτηματολόγιο. Γι' αυτό, εάν θέλουμε να είμαστε πιο σκληροί, αν θέλουμε να διευρυνθεί η σφαίρα επιρροή μα. θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τροποποιήσει ε, αυτό το ερωτηματολόγιο Δεν μπορούμε όμως να υποχρεώσουμε κάποιον ε, και ε, ακριβώς αυτό έγινε το πρόβλημα. Η κυρία Ρέγνερ το υπέδειξε. Παραδείγματος χάρη ε, τα εξαρτώμενα τέκνα, τα μέλη της οικογένειας ε, του ε, διοριστέντα επιτρόπου έχουν παραδείγματος χάρη συμμετοχές, μετοχές σε εταιρείες Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουμε μέχρι ποια, ε, μέχρι ποιο σημείο θα φτάσουμε. Για όλα τα μέλη της οικογένειας θα θέλουμε να έχουμε τέτοιες ε, πληροφορίες στην ε, Επιτροπή Γεωργίας παραδείγματος χάρη. Αν αγοράσει υποψήφιος επίτροπος 100 εκτάρια γης και θέλει να καλλιεργήσει ξέρω, καλαμπόκι όταν είναι εν ενεργεία επίτροπος. Τώρα ε, ε, υπάρχει λόγος να τροποποιηθεί η δήλωση οικονομικών συμφερόντων ή ε, να αλλάξει το χαρτοφυλάκιό του. Μόνο και μόνο επειδή θέλει να καλλιεργήσει καλαμπόκι θα πρέπει αναλογικά να δρούμε και να βλέπουμε ακριβώς τι είναι σημαντικό σε κάθε περίπτωση. Αν θέλετε να λειτουργούν όλοι υπεύθυνοι, και να αποφύγουμε τέτοια προβλήματα, ας αποφύγουμε και εμείς αυτή την αμφίβολη ε, προσέγγιση που μας προτείνεται. Το... Σε καμία περίπτωση πρέπει εμεί να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία να τροποποιήσουμε το ρετοιμοτολόγιο τι και πότε πρέπει να δηλωθεί. σε αυτές τις ακροάσεις των διοριστέντων επιτρόπων το Κοινοβούλιο ε, εξετάζει μόνο τα οικονομικά συμφέροντα αυτών. Τα ε, άλλα ζητήματα εξετάζονται από τις καθήλυν αρμόδιες επιτροπές. Είναι διαφορετικά τα ζητήματα. Ε, θα πρέπει να ξέρουμε επίσης τι γίνεται κατά τη διάρκεια της θητείας. Μπορούμε να θέσουμε ε, ε, ζητήματα επί ποιας βάσεως. Αν υπάρξουν 15 δημοσιεύματα με ανεξακρίβεται σε πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιώσει οι αρχές. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις που θα είναι ικανοποιητικέ για όλους και κυρίως σε διαθεσμικό επίπεδο, οργανικό επίπεδο, γιατί εμπλέκεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να αποφύγουμε οτιδήποτε οδηγεί σε πολιτικά παιχνίδια και σε τροφοδότηση των πολιτικών εντάσεων. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κύριος Καβαντά. Εντάχει χωρίς να μπούμε σε συζητήσεις, ε, κύριε Ζεύκα, θα συμφωνήσω με το τελευταίο σκέλος της παρέμβασής σας ε, ε, και θέλω να επιμείνω γιατί νομίζω ότι δεν εισακουστήκατε. Θα ήθελα εγώ να σας δώσω για ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Τι έχω στο μυαλό μου, τόσο ώστε να βοηθήσουμε έστω και οριακά τον συνάδελφο Ντυρά για να τελειοποιήσει την έκθεσή του. Φυσικά εγώ θεωρώ ότι είναι ήδη ε, μάλλον πλήρης η έκθεση. Τέλος πάντων, δύο είναι τα ζητήματα. Πρώτο επειδή υπάρχει υποψία συγκαταβατικής συμπεριφοράς από πλευράς του κοινού, ζητούσα ένα πληρέστερο ερωτηματολόγιο. Συμφωνώ όμως μαζί σας, πού θα σταματήσουμε, μέχρι πού θα πάμε. Είναι δύσκολο να το προσδιορίσουμε και γιατί το λέω αυτό, διότι το θέμα είναι το τωρινό ερωτηματολόγιο, όπως με τον κύριο Μπαρόζο. Εκείνο σεβάστηκε τον κανόνα της Επιτροπής. Δεν είναι καλός ο κανόνας όμως. Δεν επαρκεί. Έχουμε ε, κατά κανόνα... Ε, αυτή την περίοδο 5 έως και 7 χρόνια σε αυτή την περίοδο δεν μπορεί να υπάρξει σύγκρουση συμφερόντων ε, σε σχέση με το αξίωμα που είχε ε, ο εν λόγω επίτροπος. Αυτό, αυτά λέει ο κανόνας. Δεν είναι καλός, τροποποιήθηκε πριν από δύο χρόνια, δεν επαρκεί όμως, θα πρέπει να συμπληρωθεί. Ε, και το βλέπουμε τώρα με τον κύριο Μπαρόσο δεν μπορούμε να τον κατακρίνουμε, διότι δεν παραβίασε τον κανόνα. Απλώς δεν είναι καλός ο κανόνας. Ο ΚΟΚ, άμα σας επιτρέπει να ε, είσαστε στα αριστερά, ενώ πρέπει να πηγαίνετε στα δεξιά ή το αντίστροφο, δεν είναι καλός ο ΚΟΚ και θα υπάρξουν θύματα. Δεν είναι το, ε, το, ο υπέτειος ε, δεν είναι ο και το θέμα δεν είναι μόνο η εξακρίβωση των πληροφοριών που λαμβάνει το Κοινοβούλιο. Οι πολιτικοί αντίπαλοι ή οι φήμε στον τύπο μα ενημερώνουν προ το παρόν. Δεν έχουμε τίποτα άλλο στη διάθεσή μα και κρίνεται η μοίρα κάποιου ε, με αυτέ τι κατά προσέγγιση πληροφορίε που έχουμε. Και υπάρχει ε, μια δεύτερη υποψία που σχετίζεται με τι πράξει ε, του διοριστέντα επιτρόπου. Χωρί κανένα πολιτικό χρωματισμό, θα ήθελα μόνο να πω ότι επειδή μιλάμε για την υποψία για τον κύριο Καλνιέτε, επικρατεί λοιπόν αυτή η καχυποψία σε σχέση με τον κύριο Καλνιέτη για την μεταβίβαση ε, τίτλων ιδιοκτησία στην οικογένειά του. Αν ήμουν οραχό για να προστατεύσω τη χώρα μου, το κόμμα μου, την ε, Ισπανία, γιατί θα ηγεί σε πολύ σημαντικέ διεθνεί διαπραγματεύσει, εγώ προσωπικά θα επέλεγα να το αποδοθεί ένα διαφορετικό χαρτοφυλάκιο. Για να, για να, για να ε, ξεκαθαρίζουμε αυτά τα ζητήματα και μετά την υπόθεση Κρέσο, έχουν περάσει 28 χρόνια, ε, ε, για να ξεκαθαρίσουμε αυτά τα ζητήματα μία και έξω, για να διασκεδάσουμε οποιασδήποτε ανησυχίε ε, ανησυχίες, υποψίες υπάρχουν, νομίζω ότι θα πρέπει να επιδιώξουμε την τροποποίηση αυτού του κανόνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, δεν ζητεί κανείς τον λόγο επομένως. Σας αναφέρω ότι η προθεσμία για τις τροποποίηση αυτής της έκθεσης είναι 13 ενάτου, εάν δεν έχετε αντίρρηση. Δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια αντίρρηση, πρόταση αλλαγής αυτής της προθεσμίας, οπότε και συνεχίζουμε με το σημείο υπαριθμών 12, που είναι η συζήτηση ε, σχεδίου εκθέσεων που φορτούν. Κατά τον τρίτο χρόνο κάτι οίκοι των οποίων υπόκειται στην υποχρέωση θεώρηση διέλευση εξωτερικών και τρίτων χώρων. Και οι πίκοι αυτών των χώρων απαλλάσσουν από την υποχρέωση αυτή και συγκεκριμένα η έκθεση αυτή αφορά την Ουκρανία και τον λόγο έχει η Σύρδη κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, με μεγάλη μου χαρά να σας παρουσιάσω ε, αυτή μας την σύσταση ότι δηλαδή θεωρούμε πως ε, η Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών ε, Δικαιοσύνη και στον Υποθέσεων προτείνει σε πρώτη ανάγνωση να εγκριθεί αυτό το κείμενο ακριβώ όπω το προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θυμάμαι είχα ε, παραστεί στην στην συνάντηση κορυφή τη ε, ε, εταιρική σχέση προ Ανατολά και ο πρόεδρο Ποροσέγκο είχε αναφέρει ότι είχαμε αυτή την διαδήλωση των, έξω από το κτίριο που έλεγε ε, ότι θέλα να καταργηθεί αυτή, αυτός ο περισμός και λέγανε ότι δεν γεννήθηκα δέσμιος στη όρση διαβατηρίου και μας έλεγε ότι οι Ουκρανοί θέλαν διακαώς να υπάρξει αυτή η κατάργηση της ε, θεώρησης διαβατηρίου και ότι αξίζει ο αυτός να αμυφθεί ε, να έχει αυτό το πράγμα σαν ε, ε, αμοιβή λοιπόν για όλες αυτές τις επόδυνες μεταρρυθμίσεις που γίνονται στη χώρα. Βέβαια, όπως και στη Λουφανία έχουμε τώρα κάποιες κατηγορίες από Γερμανία και Γαλλία γιατί υπάρχουν δυσάρεστα στατιστικά στοιχεία για παράνομη μετανάστευση και για εγκληματική δραστηριότητα. όμω σύμφωνα με την εκθέση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής, ε, όλα τα προαπαιτούμενα για κατάρτιση βίζας τα πληρεί η χώρα. Οπότε σας προτείνω να έχουμε αυτές τις τέσσερι παραγράφους, τόσο ώστε να αιτιολογείται η πρότασή μας. Και έτσι λαμβάνουμε υπόψη τα συμπεράσματα τα οποία εσεί πρόεδρε ε, και, και άλλοι συνάδελφοι και υποφαινομένοι ε, είπαμε ότι ισχύουν το Σεπτέμβριο κατά την εμψυχή μας στη χώρα. Οπότε και είχαμε και επαφές με τις εκεί δικαστικές αρχές γιατί διαπιστώσαμε ότι αποδίδει το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί έχουμε αυτή την ε, συμβουλευτική υπηρεσία που βοηθά την χώρα και είπαμε Επίση, ως ε, αιτιολόγηση να ληφθεί υπόψη το πόσο έχουν προοδεύσει όσον αφορά την μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. Θα πρέπει όμως να υποστηριχθούν τα επιδεύματα της χώρας γιατί έτσι είναι δυνατόν να υπάρξει για όλες τις ε, κατηγορίες ε, της εκεί κοινωνίας ε, το κράτος δικαίου. Πολύ σημαντικό το έργο που τελείται εκεί δεδομένης της ιστορίας και της σημασίας της χώρας. Ο πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω να ζητεί κάποιο το λόγο. Α, με συγχωρείτε εσείς κύριε Φως. Μια ερώτηση κυρία Χαουταλά, αν με επιτρέπετε. ως εξής. Γνωρίζετε ποια είναι, ποιες είναι οι επιπτώσεις του Ολλανδικού όχι στο δημοψήφισμα. Μήπω Μήπως είναι παρούσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων, γιατί η ερώτησή σας μάλλον απευθύνεται σε αυτά τα όργανα. Θεωρώ ότι είναι αναπόφευκτο ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στη Συμφωνία Συνδέσεως καθώς και στην ε, ε, συνολική αυτή ε, συμφωνία βοήθειας. Αλλά δεν θα είναι θεμελιώδεις οι αλλαγές αυτές. Αν όμως κάποια χώρα μέλος, ακόμη και σε συμβουλευτικό δημοψήφισμα, απορρίψει την συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας, αυτό αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα και πρέπει να ληφθεί υπόψη. Δεν γνωρίζω βέβαια τις λεπτομέρειες των διαπραγματεύσεων. Εξ όσων γνωρίζω δεν έχει επηρεαστεί το θέμα της απελευθέρωσης των προξενικών θεωρήσεων. So, uh, thank you very much. May I say that... Ο πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Αν ε, θα θέλατε να σας πω ότι η 20 Σεπτεμβρίου είναι η υποθεσμια των καταθέσεις τροπολογιών, 12η μεσημβρινή, δεν βλέπω να uh, ενίσταται κανείς, ώστε Συνεχίζουμε με το υπαριθμό 13. Εξέταση σχεδίου γνωμοδοτήσεως για μια συνεκτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσης για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητος. Και ε, η συγκίτρια είναι η κυρία Τερέζα Κομοδίνη Κάτσα. Ζητώ συγγνώμη που σας ε, διαβίβασα την έκθεση μέσα στι θερινέ διακοπέ. Ήταν όμως οι προθεσμίε που μου είχαν επιβληθεί και ήθελα να ολοκληρωθεί η έκθεση ε, εγκαίρως. Η έκθεση συντάχθηκε λοιπόν μέσα στον Αύγουστο για να μπορέσει να αποσταλεί και στην μετάφραση. Οι σύντομε προθεσμίε, συνεχίζονται. Προσπάθησα ε, να επιτύχω μακρότερες προθεσμίες, αλλά η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών μου λένε ότι είναι μέχρι την πέμπτη της τρέχουσας εβδομάδος. Πάντως στην αρχική έκθεση και επειδή υπάρχει περιορισμός των στοιχείων που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς, δηλαδή των χαρακτήρων που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς, αλλά και επειδή περιοριζόμαστε από το πεδίο των αρμοδιοτήτων μας, λόγω των περιορισμών λοιπόν αυτών προσπάθησα να στοχεύσω την έκθεσή μου γύρω από τέσσερα ιδιαίτερα στοιχεία της αναγνώρισης των αποτελεσμάτων της ψηφιοποίησης στον τομέα CCI, να ληφθεί υπόψη η διαπραγματευτική ε, δυνατότητα δύναμη των ΜΜΕ, πειρατεία και ορθή αποζημίωση των δημιουργών. Έχουμε βέβαια εξετάσει και την γνωμοδότηση που κατέθεσε η Επιτροπή Πολιτισμού αλλά και η Επιτροπή ΙΜΚΟ. Στην Επιτροπή Πολιτισμού παρακολουθούμε και την διαδικασία των τροπολογιών που διεξάγεται τώρα και θα χρειαστεί να περιορίσουμε τις τροπολογίες μας επί της ε, γνωμοδοτήσεως μόνο βέβαια μέσα στα πλαίσια αρμοδιοτήτων της Επιτροπής μας. Έχουμε δύο συγκεκριμένες τροπολογίες που θα ήθελα να καταθέσω εγώ η ίδια. Δεν είναι τροπολογίες βέβαια για τα όσα ήδη έχουν γραφτεί. Και η πρώτη είναι, σχετίζεται μάλλον με, την, με τον ορισμό των CCI, Convergence and Competitive Instrument, εκεί γίνονται κάποιες προτάσεις να περιγράφουμε δηλαδή έναν ορισμό των CCI, είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε για ποια πράγματα μιλούμε, να γνωρίζουμε για ποιους κλάδους μιλούμε. Θα είναι όμως νομίζω επικίνδυνο να εγκρίνουμε εξαντλητικό ορισμό, γιατί ακόμα και μέσα στον χώρο αυτό των δημιουργών, εν ώψη των εξελίξεων της ψηφιοποίησης και της τεχνολογίας, νομίζω με τον τρόπο αυτό θα βλάψουμε τον τομέα περισσότερο, εάν δηλαδή περιλάβουμε έναν εξαντλητικό ρυθμό αντί για ένα γενικότερο πλαίσιο. Το δεύτερο στοιχείο που θα ήθελα να προσθέσω μέσω τροπολογίας θα ήταν να αναφερθώ στην παράνομη επιγραμμική κυκλοφορία περιεχομένου και πώς αυτή επηρεάζει το copyright. Εφόσον μέχρι τώρα έχουμε εξετάσει τα ISP και τους digital stakeholder, σαν αυτούς που παραβιάζουν ή που ενδεχομένως παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Και όχι τόσο αυτούς οι οποίοι θα προωθήσουν και θα προστατεύσουν το copyright. Θα διεξαχθούν συναντήσεις με τους ε, σκιώδης ηγητής και βεβαίως αναμένω και τις τροπολογίες σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Αν με συγχωρείτε, ο κύριος Νεγκρέσκου έχει ζητήσει το λόγο στα αγγλικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύντομη παρέμβαση. Και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αναφερθούμε στον ορισμό των CCI που γίνεται στην αρχική έκθεση. Αυτός είναι κάπως περιορισμένος, διότι αγνοεί τις νέες τάσεις που σημειώνονται στην κοινωνία, δημιουργίας δηλαδή, περιεχομένου κλπ. Θεωρώ επίσης ότι πρέπει να αναφερθούμε και στην ψηφιακή δημιουργικότητα και ψηφιακό πολιτισμό. Στην αρχική έκθεση βλέπουμε αναφορές σε αυτά και, κατά τη γνώμη, και στη γνωμοδότησή μας μάλλον αναφερόμαστε στον ψηφιακό τομέα όμως δεν προσφέρουμε χώρο για τη δυνατότητα να δημιουργηθεί ψηφιακή δημιουργικότητα και ψηφιακός πολιτισμός και πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτό. Και αναφερόμενοι στις αρμοδιότητες μας πρέπει να γίνει κάποια αναφορά και στο νομικό πλαίσιο για τους επαγγελματίες οι οποίοι εργάζονται στον τομέα αυτό και εκεί να είμαστε πολύ ακριβείς και να τους προσφέρουμε τα ίδια δικαιώματα σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα επιτρέψει το έργο μας να είναι πολύ πιο επιτυχές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λεπρόεδρος. Δεν έχω άλλον που να ζητεί το λόγο. Επειδή, η, όπως είπε μάλλον η κυρία Κομοντίνη Κατσία, η προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών είναι η 8η ενάτου στις 12 το μεσημέρι και πάλι. Ευχαριστώ λοιπόν. Ακολουθεί το άρθρο, συγγνώμη, το ε, σημείο 4 παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, REFIT σε σχέση με την πρόταση για συμβάσεις για επιγραμμικές και εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών. Σας δίνω το λόγο για 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους με την ευκαιρία. Πάντως να ευχηθώ σε όλους ε, καλό χειμώνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα τηρεί την υπόσχεσή της του Δεκεμβρίου του 2015, διότι τότε εγκρίναμε την ε, πρόταση για ιντερνετικές ε, πωλήσει ε, αγαθών και εμπορευμάτων. Και ταυτόχρονα είπαμε ότι θα μελετήσουμε και θα συλλέξουμε στοιχεία και δεδομένα για την λειτουργία των πωλήσεων γίνονται από κοντά, face to face και να εμπλακεί και το Συμβούλιο για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να ευθυγραμμίσουμε τις, ε, τους κανόνες που έχουν ε, ε, εγκριθεί. Και έχει προχωρήσει αυτή η διαδικασία και καθίσαμε λίγους μήνες γιατί συλλέξαμε στοιχεία στα πλαίσια του ευρύτερου προγράμματος REFIT, δηλαδή του προγράμματος για βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου. Αυτό είναι κάτι ευρύτερο και είπαμε ότι έχουμε εδώ έξι νομοθετήματα που αφορούν τέτοια ζητήματα καταναλωτών και λοιπά και εμπορικά ε, για παραπλανητική διαφήμιση, για ε, επισήμανση της τιμής, δικαιώματα των ε, καταναλωτών, γιατί είπαμε ότι με το νομοθέτημα αυτό είπαμε ότι ρυθμίζει το τι γίνεται όταν κανείς αγοράσει κάτι το οποίο είναι λατωματικό. Είναι ένα από τα έξι σχετικά νομοθετήματα, αλλά για να μπορέσουμε να τηρήσουμε την υπόσχεση προς εσάς ε, προσπαθήσαμε να ε, έχουμε κάποια, κάποια παραρτήματα που θα επισυνάπτονται και αυτό απλώς είναι το πρώτο πιάτο και θα ακολουθήσουν και άλλα νομοθετήματα όσον αφορά αυτού του είδους τις πωλήσει face to face. Τι γίνεται, έχουμε συνεντεύξεις. Συνεντεύξεις που είναι 23.000 σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, συν Νορβηγία, συν Ισλανδία. Επίσης ε, Μιλήσαμε 372 ε, πολιτές λιανικής και επίσης με κάποιες πολύ μικρές επιχειρήσεις και μικροεπιχειρήσεις. Οπότε δεν ήταν μόνο θέμα ποσότητος, αλλά προσπαθήσαμε να έχουμε επαφή με, πρόσωπα που εμπορεύονται ε, στην αγορά. Πολύ σημαντική είναι η μελέτη του 2015 της Επιτροφής και αφορούσε τις ε, νομικές και εμπορικές εγγύσεις. Τώρα τι άλλο ε, βρήκαμε ότι έχουμε πάνω από 3 εκατομμύρια ε, εμπόρους λιανικές και 35% αυτών ήδη σήμερα λειτουργούν ταυτοχρόνως και ιντερνετικά και επίσης όπως και σε κάποια τέτοια καταστήματα και θα πρέπει να δούμε αν θα έχουμε δύο διαφορετικά νομοθετήματα γιατί πρόκειται για εκατομμύρια ε, λιανοπολιτών οι οποίοι θα υποστούν τη συνήπωση της νομοθεσίας. Επίσης διαπιστώθηκε έχουμε 42% λιανοπολιτών τέτοιων οι οποίοι χρησιμοποιούν τέτοιου είδους ε, ε, μεθόδους face to face και έχουν πρόβλημα για διασυνορικές πωλήσει γιατί υπάρχουν, ε, υπάρχει διαφορετικό ενοχικό δίκαιο σε κάθε χώρα. Οπότε έχουμε 46% επίσης των ε, τέτοιων εμπορευμένων που χρησιμοποιούν τις ε, διατάξεις που ισχύουν για πωλήσει εξ αποστάσεως. Πολύ σημαντικό αυτό. Και επομένως υπάρχουν προβλήματα σε διασυνοριακές συναλλαγές. Σήμερα οι καταναλωτές δεν ε, συναλλάσσονται ούτε τόσο ιντερνετικά ούτε τόσο και Οπότε εδώ υπάρχουν δυνατότητε να έχουμε εκμεταλλευτεί. Για κοιτάξτε τα ποσοστά. Έχουμε 73% των καταναλωτών οι οποίοι ε, κάνουν συναλλαγές ε, υλικέ, φυσιολογικές ας πούμε, σε ένα μαγαζί. Και μόλις 11% οι οποίοι έχουν πάει σε κάποιο κατάστημα, σε κάποια έμπορο, σε κάποια άλλο κράτος μέλος από το δικό τους. Ε, Βεβαίω και υπάρχει λόγω το χαμηλό ποσοστό, γιατί όλα αυτά είναι δυνατότητες που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη. Ε, κοιτάξτε τι γίνεται με τα διαρκή αγαθά, ας πούμε έναν ε, υπολογιστή ή μια οικιακή συσκευή. Μόνο 5% των καταναλωτών έχουν ταξιδέψει σε κάποιο άλλο κράτος μέλος, ούτως ώστε να αγοράσουν τέτοια διαρκή αγαθά. Οπότε θα πρέπει να δούμε εδώ πέρα οι επιλογές πάνω για την πολιτική μας. Αυτά θα πρέπει να σας ε, αποσχολήσουν όπως και οι νομοθέτες. Πρώτα το ζήτημα είναι οι εγγύησει του νόμου. Ξέρετε το Δεκέμβριο του 2015 τι προτάσεις υπήρχαν. Ότι θα πρέπει να ε, πάμε σε πλήρη εναρμόνιση. Και είπαμε ότι για οτιδήποτε είδους ελάττωμα να προβλέπεται εγγύηση διετής. Πλήρης εγγύηση, ούτως ώστε να μπορεί κάποιος να ζητήσει αποκατάσταση ή ε, αποζημίωση. Και οι εμπορευόμενοι, τους οποίους ρωτήσαμε, είπαν ότι τέτοιου είδους πλήρης εναρμόνιση ε, είπαν ότι αυτό θα ήταν το κόστος. Αλλά πολύ περισσότεροι ε, είπαν το ίδιο όσον αφορά κάποιους, ας πούμε, όπως Σουηδία, Φινλανδία ε, και κάτω χώρες. Γιατί εκεί υπάρχει μεγαλύτερη, μακρότερη περίπτωση εγγύησεως. Επίσης, επίσης ε, ρωτήσαμε τις επιχειρήσεις πώς τους φαίνεται ε, η συνέπεια της διατάξεως σύμφωνα με την οποία φέρουν ευθύνη κατά όλη την διετία. μεγάλο ποσοστό, ακόμη περισσότεροι από όσου βλέπετε εδώ στο κείμενο, γιατί είπαμε ότι επεξεργαστήκαμε αυτά τα δεδομένα και θα δείτε το τελικό κείμενο τέλος Σεπτεμβρίου, οπότε ακόμα περισσότεροι από το 60% είπαν ότι αν γίνει τέτοιου είδους ε, εναρμόνιση ε, δεν θα οδηγούσε σε κάποια επιβάρυνση. Πολύ σημαντικό αυτό για τους καταναλωτές ούτως ώστε να καλυφθεί η περίπτωση ε, της του σχετικού δικαιωμάτους. Τώρα όσον αφορά την ιεραρχίζει των ε, ενδίκων μέσων, των μέσων τελευταίων που υπάρχουν για αποκατάσταση και είπαμε τι γίνεται για, ε, σχετικά με επισκευή για αντικατάσταση. Και αν δεν είναι δυνατόν να έχουμε κάποιο είδου μείωση του τιμήματος. 51% των καταναλωτών είπαν ότι δεν ζητούν λύση της συμβάσεως ευθύς αμέσως και πρώτα προσπαθούν να πετύχουν την επισκευή ή την αντικατάσταση του ερωτηματικού αγαθού. Αυτό ισχύει και στις χώρες που σήμερα έχουμε δευτερογενές δίκαιο που αφορά την ελεύθερη επιλογή ε, της, της αποκατάστασης. Δηλαδή Κροατία, Λιθουανία και Ελλάδα. Και εκεί συμφωνούν ε, όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία όμως θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά και θεωρήσαμε ότι έπρεπε να σας τα αναφέρουμε τώρα. Τελευταίο αλλά σημαντικό, η επιλογή όσον αφορά ε, την κατάρριξη της ε, υπόσχεσης, της συγγνώμη της καταναλωτή να μπορέσει, να, να υποχρεούται να καταγγείλει ένα πρόβλημα μέσα στο δίμηνο. Αυτό το οποίο διαπιστώθηκε ήταν ότι αφενός Έχουμε πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις οι οποίες είπαν ότι αν αρθεί αυτή η υποχρέωση δεν θα ε, φέρνουν κάποιο κόστος, κάποια ζημία ή θα είναι πολύ μικρό το κόστος. Σας επισημαίνω επίσης ότι γνωρίζουμε από μελέτες ότι οι καταναλωτές γενικά είναι πολύ δυναμικοί σε αυτό το μέτωπο και οι περισσότεροι επισημαίνουν το ελάττωμα είτε αμέσως είτε τις αμέσως επόμενες πρώτες μέρες της ε, αγοράς του αγαθού. Οπότε θα πρέπει να δούμε κατά πόσο χρειάζεται να συνεχίσει να ισχύει αυτός ο κανόνας. Προσπάθησα να είμαι πάρα πολύ σύντομη, αλλά βέβαια πολύ περισσότερο μπορούσαμε να πούμε, αλλά να σας τα πω εάν χρειαστεί και με ρωτήσετε σχετικά. Do I understand that Mr. Le asks for the floor? Κατάλαβα καλά, κύριε Λεπρετών, θέλει το λόγο. Καλά, η κυρία Χατάλα τότε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση, διότι παρουσιάζω το της πρότασης σε σχέση με ε, τις ε, συμβάσεις ε, πολίσεων για αυτά αγαθά. Θα ήθελα κάποια ε, πρώτα ζητήματα να τα γύρω ήδη. Είναι σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, να υπάρχει συνοχή και συνέπεια ε, ομοιομορφία κανόν ανάμεσα σε όλες τις κατηγορίες πωλήσεων επιγραμμικών ε, ή όχι. αξιέπαινος αυτός ο στόχος που έχετε από την άλλη πλευρά και νομίζω ότι έχετε πλήρη επίγνωση κατάσταση από τις συζητήσεις που είχατε με τα κράτη-μέλη, ότι λοιπόν, εάν επιλέξουμε ε, την ευθυγράμμιση των κανόνων, το αποτέλεσμα θα είναι ε, να υποβαστούν τα πρότυπα προστασίας των κατανοητών σε κάποια κράτη-μέλη στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Φινλανδία, στη Σουηδία, πώς να εξηγήσουμε στους καταναλωτές ότι ξαφνικά θα υπάρχει αυτός ο περιορισμός για τη διετή περίοδο, ε, για την ε, νομική εγγύηση που υπάρχει, ο περιορισμός δηλαδή στα δύο χρόνια. Μην ξεχνάτε επίσης ότι υπάρχει το θέμα της διάρκειας ε, του κύκλου ζωής των προϊόντων. Δεν είναι θετικό αυτό το σημάδι. Ότι δηλαδή ε, ο, ο αναμενόμενος κύκλος ζωής των προϊόντων τελικά είναι αυτή η διετής περίοδος που εμείς εγγυούμαστε. Είναι ένα δίλημα το οποίο είχαμε από τα πρώτα βήματα της ε, νομοθεσίας ε, για τις πωλήσει. Επειδή όμως είμαι διαλύτρια, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή την ευθυγράμμιση δεν μπορούμε να την κάνουμε προς τα πάνω στο ανώτερο επίπεδο προστασίας, παραδείγματος χάρη για αυτή την περίοδο προστασίας των καταναλωτών. Γιατί εμείς εδώ στο Κοινοβουλίο θα περιέλθουμε σε δινή θέση. Πώς θα εξηγήσουμε στους καταναλωτές ότι έφνης θα απολέσουν δικαιώματα που με μεγάλη χαρά έχουν κατοχυρωθεί. Ε, έχουν δει να κατοχυρώνονται. Ε, και ότι ε, εντάξει παρότι θα προέρχεται αυτό από διασυνοριακές πωλήσει, νομίζω ότι θα πρέπει να <coughs> επιδιώξουμε, όπως σωστά είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνοχή και να επιδιώξουμε ευθυγράμμιση στο ανώτατο δυνατό επίπεδο προστασίας. Για να δούμε τι θα καταφέρουμε. Θέλει εντάχει να απαντήσει ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρο. Ευχαριστούμε κυρία Χάουταλα, θεμητό το ερώτημά σας και γράφτε πλήρως τη συζήτηση που κάνουμε. Φυσικά θα μπορούσαμε να το φανταστούμε και φυσικά το έχουμε θέσει ως ζήτημα διότι το ζητούν και ενός καταναλωτών. Το πρόβλημα είναι πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει ένα διτό στόχο μέσω της πρότασης. Αφενός να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των κατάλληλων σε διασυνοριακές ε, πωλήσει, αλλά και εθνικές, απ' την άλλη δε να διευκολύνει και τις επιχειρήσεις να πολλούν δηλαδή διασυνοριακά αλλά και ε, στο εσωτερικό της χώρας ε, τα προϊόντα τους. Και ιδιαίτερη εστίαση επί των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως είπε συνάδελφος με Φρέντι. Επειδή έχουμε λοιπόν αυτό το διπλό στόχο και ο απότερος στόχος είναι αξιοποίηση του δυναμικού ε, του ηλεκτρονικού εμπορίου ως κινητήριου δύναμης ε, του εμπορίου γενικότερα. Πρωτού καταθέσουμε την πρόταση στη δημόσια διαβούλευση που έγινε μεταξύ το 2015, προσπαθήσαμε όπως σε πολλού τομεί να βρούμε τη μέση οδό. Αν επιδιώξουμε το ανώτατο επίπεδο προστασίας, φυσικά θα υλοποιήσουμε το στόχο τη ενίσχυση τη εμπιστοσύνη των καταναλωτών, διότι καλύτερα δεν θα γίνεται, όμως δεν θα ενθαρρύνουμε τι επιχειρήσει, ιδίω δε τις μικρομέσαίε να πολλούν διασυνοριακά. Γι' αυτό υπάρχει ένα υψηλότερο επίπεδο προστασία στην πρότασή μας, σχεδόν σε όλα τα σημεία. Υπερβαίνουμε τα προβλεπόμενα στην κείμενη οδηγία. Παρατείνουμε την περίοδο από 6 σε 2 χρόνια για το βάρος της απόδειξης. Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο που μπορεί να έχει ένα κράτος μέλος. Οπότε πιστεύω ότι στο επίπεδο που είμαστε ε, επιτυγχάνουμε ταυτόχρονα και τους δύο στόχους. Ευχαριστούμε. Δεν ζητά κάποιο άλλο το λόγο. Οπότε... Θέλω να ευχαριστήσω και τους δύο εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρουσίαση. Και από αγαπητά μέλη, επιτρέψτε μου. Ε, προβλέψαμε στι 5 παρατέταρτο να ψηφίσουμε. Θα ήθελα λοιπόν ευθύ αμέσω να περάσουμε στην ψηφοφορία και να συνεχίσουμε ε, με όλα τα υπόλοιπα σημεία. Παρακαλώ, ετοιμάστε τι κάρτε ψηφοφορία. Thank you. Mrs. Regner, uh, Κυρία Ρέγνερ, πρόεδρε, σημειώστε παρακαλώ ότι ξέχασα την κάρτα μου και θα σηκώνω το χέρι. αυτό είναι στις καλές παραδόσεις της Επιτροπής μας. Ας αρχίσουμε. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. πέτει 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13. Έμπλη 18, υπέρ. 3. In favor. Πέτησε 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έκον 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Για την έκον 1. Uh, rejected. Uh, then ample, ample two. Ample zero Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πέτει ένα υπέρ. Ample ε, 3, sorry, Ample 3 in Ample 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έκον 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 12. Έκον 3, όχι έμπλη 12, έκον 3 υπέρ, κατά, αποχές, α, απορρίπτεται. Η πρώτη συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έκον 20 θα λέω. Ναι, ναι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 5 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 39 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές Επαλήθευση παρακαλώ. Yes. Adopted. Uh, yeah, it's it's, adopted. adopted. Uh, Εγκρίθηκε. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 49 κάποιος λέει όχι. Απερίφθη. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και αυτό 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 υπέρ κατά παρακαλώ επαλήθευση ηλεκτρονική επαλήθευση Εγκρίνεται αυτό. Κύριε Πρόεδρε, η κυρία Χάουταλα. ω εισηγήτρια. Εάν 57 και 55 έχουν ακριβώς την ίδια πλειοψηφία νομίζω θεωρήθηκε ότι απορρίφθηκαν αλλά δεν είμαι πεπισμένη βλέποντας τώρα την ηλεκτρονική ψηφοφορία της 58 με την άδειά σας να ελέγξουμε πάλι τις 55 και 57 η κυρία Ρέγνερ Στην τελευταία δεν είπατε εγκρίνεται, εγώ όμως ψήφισα κατά. Ο κ. Βιέφκα ψήφισε υπέρ όμως. Uh, Έχει καλώσει 58. Θέλετε όμως τώρα να επαληθεύσουμε την 55 και 57. Συμφωνείτε κυρία Χάουταλα, αυτό ζητήσατε. Ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν 55 απορρίπτεται. Θέλετε και την 57. Όχι, νομίζω ότι είχατε απολύτως δίκαιο. Άλλωστε δεν είχα και κανένα λόγο να υποπτευθώ το αντίθετο. Καλά κάνετε όμως και με ελέγχετε γιατί μετά τις διακοπές αντιλαμβάνεστε Ακόμα δεν είμαι ε, πλήρως εδώ. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά. Αρχές. Απορρίπτεται. 23 της Οικονομικής Επιτροπής. Φαίνεται πως υπάρχει προφορική τροπολογία του εισηγητού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αναφορές 7 υπέρ. Κατά. Α, όλες μαζί λέτε. Από την 7 όλες μαζί μέχρι την έμπλ 25. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται όλες αυτές.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 αποχές απορρίπτεται. Το ίδιο ισχύει για την υπαριθμόν 6. 7 υπέρ. Υπέρ. Πάντα. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έκον α υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έκον ε, β υπέρ Κατά. Παρακαλώ επαλήθευση για τούτην εδώ. Έκον Β. Εγκρίνεται, λέει ο πρόεδρος. Έκον σε υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται αυτή. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Το σχέδιο στο σύνολό της, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια, κυρία Χάουταλα. Θα συνεχίσουμε με την άδειά σα. με το υπαριθμό 17 ανταλλαγή απόψεων για τη γενική αναθεώρηση των κοινοβουλευτικών κανόνων με εισηγητή εμένα προσωπικά. Έχω να πω το εξή. Η Επιτροπή μας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη γενική αναθεώρηση των κανόνων, του κανονισμού δηλαδή του Κοινοβουλίου, ιδίω λόγω των οριζοντίων αρμοδιοτήτων της σε ζητήματα όπως διαπιστευ... Διαπιστευ... Δια... επαλήθευση εντολής, ασυλίες κλπ. Δεύτερο, την θέση ισχύ της νέας διοργανικής συμφωνίας για την βελτίωση της νομοθεσίας. Αυτή καθιστά αναπόφευκτη την ενημέρωση των υφισταμένων κανονισμών ή την εισαγωγή νέων. Πρόκειται για χώρο όπου έχει γενική αρμοδιότητα η νομική επιτροπή και γι' αυτό έχει και κάθε ενδιαφέρον να ακουστεί η φωνή της. Η ομάδα εργασίας της ΑΦΚΟ απέδωσε ικανοποιητικό έργο. Στη γνωμοδότησή μου θα το επιβεβαιώσω αυτό και όπου αυτό είναι αναγκαίο θα προτείνω και άλλες βελτιώσεις. Μεταξύ άλλων, θεωρώ ότι δύο θέματα αξίζουν να εξεταστούν, δηλαδή ασυλίες και νομικές βάσεις. Σε ό,τι αφορά τις ασυλίες, κοινοβουλευτικές ασυλίες. Συνολικά η νέα προσέγγιση αντιμετωπίζει ορθά τις ανάγκες της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Υπό το νέο σύστημα πάντως, οι εκθέσεις για την κοινοβουλευτική ασυλία θα τίθεται για ψηφοφορία μόνο υπόψη της Ολομέλειας εφόσον τον ενδιαφερόμενο μέλος ή μια πολιτική ομάδα το ζητήσουν. Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ο προτινόμενος μηχανισμός θα επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο βουλευτή ή στον, ε, στην ομάδα της ή την ομάδα του να αντιδρά στην έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων μέσω ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε έντονη προβολή στη δημοσιότητα με ενδεχομένω αρνητικέ επιπτώσεις κάποιων περιπτώσεων. Θα πρέπει να διατηρηθεί η ψήφος στην Ολομέλεια για κάθε αίτηση κοινοβουλευτική ασυλίας για όλους τους βουλευτές. Εκτός αυτού, επειδή οι εκθέσεις αυτές έχουν σημαντικές νομικές επιπτώσεις και ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο προσφυγών σε εθνικά ή και ευρωπαϊκά δικαστήρια, θα πρέπει να στηρίζονται και σε ψήφο της Ολομέλειας. Ιδάλλως, εκτίθεται το Κοινοβούλιο σε ενδεχόμενες νομικές προσφυγές. Δεύτερον, νομικές βάσεις. Στο προσωρινό κείμενο που εγκρίθηκε σε επίπεδο ομάδας εργασίας, οι τροποποίησει για το άρθρο 63 για εκ νέου παραπομπή στο Κοινοβούλιο υπάγονται στην ισχύ του άρθρου 25 της Διαθεσμικής Συμφωνίας ό,τι αφορά τις νομικές βάσεις. Ιδίως το άρθρο 63 παράγραφος 2 τροποποιείται με την έννοια ότι μετά από την ανταλλαγή απόψεων στην οποία γίνεται αναφορά στο άρθρο 25 της Διαθεσμικής Συμφωνίας, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, μετά από αίτηση της αρμόδιας επιτροπής, θα ζητεί από το Συμβούλιο να παραπέμπει εκ νέου στο Κοινοβούλιο σχέδιο νομοθετήματος, εφόσον Κοινοβούλιο ή Συμβούλιο προτίθεται να τροποποιήσουν τη νομική βάση που έχει εγκριθεί στην πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Με το αποτέλεσμα να μην ισχύει πλέον η τακτική νομοθετική διαδικασία. Ατυχώς, τέτοιες προτάσεις έχουν κάποιες ε, επιπτώσεις ως εξής. Γενικά, το άρθρο 63 δεν φαίνεται να είναι ιδεώδες ή πάντως και το μοναδικό μέσον για την εφαρμογή αυτού του τμήματος της Διαθεσμικής Συμφωνίας. Η παράγραφος 25 της συμφωνίας αυτής ζητεί από τα τρία θεσμικά όργανα να ανταλλάσσουν απόψεις και όχι να ανανεώνουν τις παραπομπές των νομοθετικών προτάσεων. Τέτοια επέκταση είναι δυνατή, δεν απορρέει όμως ευθέως από τη νέα διαθεσμική συμφωνία. Ίσως χρειάζεται επικαιροποιημένη διαδικασία του άρθρου 39 για την βελτιωμένη εφαρμογή της Διαθεσμικής Συμφωνίας. Δεύτερο, νέος, ε, το νέο άρθρο 63 παράγραφος 1α επιβάλλει την υποχρέωση στα άλλα θεσμικά όργανα όσον αφορά τους δικούς τους εσωτερικούς κανονισμούς. Κάτι το οποίο δεν είναι δυνατόν να γίνει για τον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου που εξορισμού δεν μπορεί παρά να καλύψει μονάχα την εσωτερική οργάνωση του Κοινοβουλίου. Τρίτο, σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Γιούρη, δεν υπάρχει καμιά διασφάλιση ότι θα διατηρηθεί ο ρόλος της. Η νέα διάταξη του άρθρου 63 εν α δεν λέει ποιος θα είναι ο εκπρόσωπος του Πρόεδρου. Εν τέλει, η συμπερίληψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παράγραφο 2 του άρθρου 63 παραβιάζει τη λογική του άρθρου που διακρίνει τις προτάσεις που γίνονται προς την Επιτροπή από αυτούς που γίνονται προς το Συμβούλιο. Όπως είπατε, προτίθεται καμία τροπολογία για το άρθρο 39, για τις νομικές βάσεις, για να προσαρμοστεί αυτό στη νέα διαθεσμική συμφωνία και ταυτόχρονα τροπολογία στο άρθρο 39 παράγραφος 3 προτείνεται ώστε η νομική επιτροπή να μπορεί να συζητεί θέματα ανα πάσα, διαδικασία, ανα πάσα συγγνώμη, φάση της νομοθετικής διαδικασίας ακόμη και εάν το Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει την θέση του όπως στην περίπτωση του άρθρου 63. Ίσως χρειάζεται μια πιο συντονισμένη προσέγγιση με την έννοια ότι θα προταθούν τροποποιήσεις και στο άρθρο 39 και στο άρθρο 63. Εγώ στην γνωμοδότησή μου θα περιλάβω όλα αυτά τα θέματα. Την δε γνωμοδότηση αυτή θα ήθελα να την παρουσιάσω στην επόμενη συνεδρίαση. Και ευχαρίστω θα ακούσω τις απόψεις σα για το θέμα αυτό. Εσείς παρακαλώ κύριε Σβιεύκα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ήταν πάρα πολύ πλήρης η ενημέρωση που κάνατε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Ό,τι τροποποίηση γίνει στον οργανισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πολύ σημαντικό για το έργο μας. Ειλικρινά σα λέω ότι συμμερίζομαι τα όσα σα προκαλούν δισταγμού και προβληματισμό όσον αφορά την ασυλία και τι ε, μελετώμενε ε, μεταβολέ θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να κάνουμε ό,τι μπορούμε, τόσο ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τίποτε δεν θα αλλάξει. Υπάρχει μια διαδικασία η οποία ισχύει για μα, η οποία είναι μια διαδικασία παγιωμένη και δοκιμασμένη και παρέχει κάποιε εγγυήσει. Αλλά επίση δίνει και το περιθώριο, τόσο ώστε να συζητηθούν όλα τα θέματα τη ε, ασυλία και παρέχονται εγγυήσει ότι υπάρχει ε, πλήρης ε, συμμετοχή του κάθε φορά εμπλεκομένου. Οπότε θα πρέπει να δούμε το ότι οποιαδήποτε τροποποίηση είναι κάτι που δεν ωφελεί, δεν εξυπηρετεί. Τα είπα και στον κύριο Βίλαντ, ο οποίος έχει αναλάβει σαν εργασία το θέμα. Του εξήγησα ε, όλες μου τις επιφυλάξεις και Ελπίζω, γιατί μίλησα και με την κυρία Χίμνερ, ότι, ότι θα μπορέσουμε να αποφύγουμε ατυχείς ρυθμίσεις και τροποποίησεις. Ευτυχώς έχουμε και τον κύριο Κόρμπετ. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Πάντως συμφωνώ 100% πρόεδρε με τα όσα είπες. Ελπίζω ότι θα προωθήσει όπω πρέπει τις θέσεις μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος και το λόγο στην κυρία Ρέγνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα αναφερθώ και εγώ στι ασυλίε, όπου νομίζω θα πρέπει και ανεπισήμως να συνομιλήσουμε τον Ρίτσαρντ Κόρμπετ Η πρόθεσή εξακολουθεί να είναι να διαμορφώσουμε με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο τις εργασίες της, της κοινοβουλευτικής ε, συνελεύσεως της Ολομέλειας. Αυτό έχει σημασία. Εάν τώρα εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τις ε, αιτήσεις κοινοβουλευτικής, ε, δηλαδή τις κοινοβουλευτικής ασυλίας, ε, έχει αποδώσει η διαδικασία αυτή ως τώρα. Ούτε θεωρώ ότι είναι καμιά μεγάλη, μεγάλη επιβάρυνση της Ολομέλειας οι ψηφοφορίες για τις αιτήσεις άψεως κοινοβουλευτικής ασυλίας. Θεωρώ λοιπόν ότι η διαδικασία έχει αποδείξει την αξία της. Νομίζω να προτείνουμε ή να προσπαθήσουμε να διαλύσουμε τις αμφιβολίες αυτές και να μάθουμε και ιδιαίτερα γιατί προβάλλουν αυτήν την αιτιολόγηση. Συμφωνώ και με τον κύριο Γεύκα. Ο πρόεδρος, ε, ευχαριστώ. Άλλος συνάδελφος δεν έχει ζητήσει το λόγο. Σας ευχαριστώ για την ανταλλαγή απόψεων και θα συνεχίσουμε με το 18 εξέταση εκθέσεως για διαδικασίες αφαιρεγγιότητας και διαχειριστές των διαδικασιών αφαιρεγγιότητας. Έχει το λόγο αγαπητέ κύριε Ζιβιεύκα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος διότι όπως ε, θα θυμάστε λίγο πριν τις ε, διακοπές εξαντλητικά είχαμε διεξέλθει το θέμα. Απλώς σας το υπενθυμίζω. Στα παρατήματα α και β θέλουμε να επιφέρουμε κάποιες τροποποίησεις όσον αφορά τις ε, πτωχευτικές ε, διαδικασίες και όσον αφορά τους νομικούς που ασχολούνται με την πτώχευση. Άρα, θα τροποποιηθεί ο σχετικός κανονισμός. Και θα πρέπει να δούμε πώς θα ρυθμίσουμε το σύνταγμά μας ε, για να είναι στο ίδιο τους με αυτές τις ε, αλλαγές. Ευρωπαϊκό Επιτροπή και το Σύνταγμα θα πρέπει επομένω να αλλάξουμε και το παράδειγμα Α και Β για την πάυση πληρωμών, την πτώχευση κλπ. Όλ, με όλα αυτά, ε, όλα αυτά μάλλον τα γνωστή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει περάσει το και από το Κοινοβούλιο της χώρας μας, οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύνταξε ένα σχέδιο κειμένου. Αυτό και τώρα ε, σχολιάζω στο σχέδιο κειμένου το δικό μου. Άρα να μην σας εκπλήξει εάν προτείνω να περάσει η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής χωρίς δικές μας τροπολογίες για τυπικούς λόγους. Ε, βέβαια, όποιο θέλει να υποβάλει κάποια τροπολογία, 9 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι είναι η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αυτών των τροπολογιών. Ο πρόεδρο. Δεν βλέπω να ζητεί κάποιο το λόγο. Συνεχίζουμε τώρα. Εγώ δεν έχει κάποιο να πει τίποτα. Έχουμε 20, 21 και 22. Εν προκειμένου η συγκήτρια είναι η κυρία Φεράρα. Όμως, ζητή συγγνώμη γιατί δεν μπόρεσε να παραστεί. If, if it is confirmed that there are uh, no objections raised against the three files. Εάν δεν υπάρχει κάποια ένσταση σχετικά, τότε θα θεωρήσουμε ότι κλείνει το θέμα συζήτησης αυτών των τριών θεμάτων. Οπότε, θεωρούμε ότι έληξαν τα τρία αυτά ζητήματα της σημερινής διάταξης. Και... Ε, Uh, you uh, uh, Όσον αφορά τώρα το θέμα υπαριθμών 23, έχετε λάβει ένα σχετικό σημείωμα αφορά την επικουρικότητα. ο κύριος Χρυσόγονος δυστυχώς δεν παρίσταται, γιατί ο κύριος Χρυσόγονος είναι ο εισηγητής. by point 20. Άρα, θα πάμε στο 24. Το 24 απαιτεί συζήτηση και κλεισμένων. Οπότε παρακαλώ όλοι οι οποίοι δεν δικαιούνται να παρίστανται να αποχωρήσουν. Thank you.